Good morning, everyone. I invite you to start the working day in our committee. I hope... Μέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε. Ελπίζω όλοι να είστε πανέτοιμοι και ακμαίοι για να ξεκινήσουμε. Αν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις ε, για την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να την εγκρίνουμε. Διερμηνία παρέχεται σε 21 γλώσσες. Ο συνήθως ε, τα έγγραφα είναι διαθέσιμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικά και υπάρχει αναμετάδοση από το διαδίκτυο. Σα στείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τι συστάσει των συντονιστών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, τι εγκρίνουμε. Έχετε λάβει και τα πρακτικά της συνεδρίασης της 20 και 21ης Μαρτίου. Οπότε και πάλι αν δεν υποβληθούν ε, παρατηρήσεις ενστάσεις ε, θεωρούνται εγκριθέντα. Το πρώτο σημείο της ημερήσης διάταξης, το κύριο σημείο, είναι η ενημέρωση για τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις Υπάρχει πρόβλημα μήπως με τη διερμηνία. Όχι, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει διερμηνία καν. Σε ποια γλώσσα, γαλλικά. Θα φροντίσουμε να διορθωθεί το πρόβλημα. Ελπίζω να επιληφθεί ο τεχνικός. Uh, so, regarding the... τριμερής ε, διάλογος για τις, τρέχου, για διοργανικές διαπραγματεύσεις. Έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος. Ε, είχαμε μια ανταλλαγή πληροφοριών με εκπροσώπους και του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα μείζωνα πολιτικά ζητήματα που γύρει αυτό το πακέτο για την κυκλική οικονομία, αυτή η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Η Συζητήσει περιστράφηκαν γύρω από τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 17 η Μαρτίου. Και κάποιε τροπολογίες που υποβλήθηκαν αμέσω μετά. Διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για κρίσιμα θέματα του πακέτου υπάρχουν ακόμη, όπως ε, τους στόχους για την ανακύκλωση και τους υγειονομικούς χώρους ταφής και τις αποκλείσει εξαιρέσει από την υλοποίηση των στόχων, απόβλητα τροφίμων και μέθοδος υπολογισμού. Παρά τις διαφορές όμως, οι συζητήσεις έγιναν σε επικοδομητικό πνεύμα και αποφασίστηκε να χορηγηθούν κάποιες εξαιρεσει από το πεδίο εφαρμογή στην ιεραρχία των, τροφί, των απορριμμάτων, Και ε, επόμενος ε, διάλογος, ε, διαμερής τρίλογος, ε, έχει προβλεφθεί για τις 26 Ιουνίου. Άλλα θέματα αφορούν τα υποπροϊόντα και την τελική κατάληξη των απορριμμάτων. Αυτά ως προς τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της διοργανικής. Περνάμε στην επόμενη έκθεση κυρίας Γκούτελαντ για την ενεργειακή απόδοση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιούτε Γκούτελαν, την εισηγητριά μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους, τους παρόντες τουλάχιστον. Χαίρομαι ιδιαίτερο που μπορώ να σας παρουσιάσω την ε, γνωμοδότησή μου για την ενεργειακή απόδοση σήμερα. Γιατί κατά τη γνώμη μου μόνο με καλύτερη αξιοποίηση των ιδίων πόρων και ξυπνότερες λύσεις των αγορών έχουμε τεράστιο δυναμικό για να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση και να πραγματοποιήσουμε σημαντικά βήματα προς μια βιώσιμη κοινωνία. Αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος. Μάλιστα το αυτή η πρωτοβουλία υπάρχει από το 2012, αλλά εξαιτία ε, κάποιων ρυθμιστικών αδυναμιών και προβλημάτων τη αγορά δεν έχουμε αξιοποιήσει το έπαρκο την ενεργειακή μα απόδοση, το δυναμικό τη ενεργειακή απόδοση. Με την αναθεώρηση αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε την κατάσταση αισθητά και γι' αυτό θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία ώστε να γίνει η ενεργειακή απόδοση κατάλληλη για το σκοπό που έχει θεσπιστεί. Η βελτίωση της απόδοσης ε, της ενεργειακής θα ενδυναμώσει την Ευρώπη και θα εξασφαλίσει ε, τον ηγετικό του ρόλο στη μετάβαση προς μια ε, κοινωνία που θα ξεπεί αποτελεσματικά τους σπόρους. Επίσης, οι επενδύσεις στον τομέα αυτό θα δημιουργήσει ε, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, έως και εκατομμύρια θέσεις απασχόληση ανάλογα με τις φιλοδοξίες μας, γιατί θα δημιουργήσει ασφάλεια, δικαίου ε, και βεβαιότητα για τις εταιρείε που θέλουν να επενδύσουν. Γιατί από το 2012 η κατανάλωση ενεργειακή έχει μειωθεί, ενώ το ΑΕΠ αυξάνεται στην Ευρώπη. Οπότε ήδη λαμβάνει η χώρα αυτή η αποσύνδεση. Είναι σαφώς, σαφές ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης συμβάλλουν ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται και στην έκθεση και στόχο έχουν να δώσουν μια όθηση στην απασχόληση με τη σωστή χρηματοδότηση και τις κατάλληλες επενδύσεις. Έχουν δείξει μελέτες ότι είναι δυνατή μια αισθητή αύξηση της απασχόλησης. Όλα, παραλαμβάνω, εξαρτώνται από το βαθμό φιλοδοξίας μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ 450.000 έως και 5 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης και ε, στόχοι υψηλής ενεργειακής απόδοσης θα αποφέρουν ε, καρπούς ε, και θα βελτιώσουν και την υγεία των πολιτών, σώζοντας χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Παίρνουμε λοιπόν την ευθύνη να βελτιώσουμε την κατάσταση για εκατομμύρια συμπολίτε μα, που υποφέρουν από την ενεργειακή ένδυα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σωστό επιμερισμό προσπαθειών ε, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την ενεργειακή ένδυα και να μειώσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας των οικοκυριών. Η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης ε, θα οδηγήσει στον περιορισμό της ρήπανσης και των αναποτελεσματικών πρακτικών, ενώ θα μειώνει και την ενεργειακή μας εξάρτηση και θα βελτιώνει την ενεργειακή μας ασφάλεια. Θα μειώσουμε έτσι τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων και στην περίοδο 2021-2030 η μείωση στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων θα μας εξοικονομήσουν 288 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους, η γνωμοδότησή μας προτείνει δεσμευτικούς στόχους 40% για το 2030 σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση. Θέτουμε εδώ τα θεμέλια για το μέλλον μας και η μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι ο στόχος του 40% είναι μακροπρόθεσμα και ο πλέον ε, αποδοτικός από άποψη τους ωφέλους και τα κρατημέρη μπορούν να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Γι' αυτό και προτείνουμε δεσμευτικούς εθνικού ε, εθνικούς στόχους για να κλείσουν τα παραθυράκια του άρθρου 7. Έτσι θα μεγιστοποιηθεί το δυναμικό βελτίωσης και σε εθνικό επίπεδο και θα αυξηθεί η προβλεψιμότητα και η βεβαιότητα ε, για τους επενδυτές, κάτι που σήμερα λείπει. Επίσης προτείνουμε υποχρεώσεις για την ανακαίνιση των δημοσίων κτηρίων ε, του άρθρου 5 παρατείνεται, επεκτείνεται για να καλύψει όλους τους δημόσιους φορείς. Τα κτίρια έχουν ιδιαίτερα μεγάλο δυναμικό βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Γι' αυτό και θα πρέπει να επισημάνω αυτό το θέμα όσο γίνεται. Μάλιστα όλες αυτές οι θέσεις ήδη επιβεβαιώθηκαν και υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάλιστα πρόσφατα, πριν από μόλις ένα χρόνο, είχαμε αυτή την ε, επιβεβαίωση. Ε, έχουμε και τη Συμφωνία του Παρίσιου, που ε, κάνει πιο ισχυρό το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της. Δεν μπορούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατρελώνουμε τη θέση μας και μετά να επαναχωρούμε όταν εκπονούμε νομοθετικές προτάσεις. Να μην ξεχνούμε και την υπόλοιψή μας και το κύρος μας. Και δύο λόγια για τους έξυπνους μετρητές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι αυτοί οι έξυπνοι μετρητές έχουν καλό δυναμικό και φυσικά θα πρέπει να είναι αναλογικό το όφελός τους, απόψη τους, ε, ή δεν να ζητηθούν άλλες πιο αποτελεσματικές λύσεις. Επίσης, στις πολυκατοικίες ε, όταν υπάρχει ένας κεντρικός λάβητας υπάρχει ένα πρόβλημα. Ε, ειδικά όταν περιλαμβάνεται στα μηνιαία κοινόχρηστα και η αλλαγή της ε, δομής θα ήταν πολύ δαπανηρή. Έτσι ίσως δημιουργηθούν ε, ε, νέες μορφές ενεργειακής ένδυας όταν οι ένικοι προτιμούν να κλείσουν τη θέρμανση για να μειώνεται το ενίκιο τους που περιλαμβάνει και το θέμα αυτό. Δεν θα πρέπει να ενισχύουμε τέτοιες πρακτικές, γιατί καλύτερα θα ήταν να δώσουμε προτεραιότητα σε άλλου είδους βελτιώσεις στην κτηριακή ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει να αναζητούνται πάντα καλύτερες ε, λύσεις από άποψη κόστους ωφέλους. Στην γνωμοδότησή μας, φυσικά, ε, αναγνωρίζουμε ότι η αρμόδια καθήλη επιτροπή είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας, εμείς απλώς συντάσσουμε εκνομοδότηση Παρ' όλα αυτά θέλω συνεργασία και με τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες και να μην ξεχνάτε και την προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών που λήγει στις 14 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γκούτελαντ. Ε, πάρα πολύ ευχάριστα τα νέα και πρέπει να προωθήσουμε την έκθεση γρήγορα. Ο κύριος Μπέλετ, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναφερθώ στον Τραμπ, ο οποίος αποσύρεται από το Παρίσι, είναι θλιβερό και βλακώδες. Τέλο πάντων έτσι είναι, αλλά δεν αλλάζει την ανάγκη εμείς να συνεχίσουμε. Να επενδύουμε σε ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτούς τους κλάδους που έχουν τις περισσότερες δυνατότητες, ε, δηλαδή τα κτίρια. Και επιτρέψατε μου να πω ως σκιώδης εισηγητής ε, για το ΙΤΙΕΣ ε, να προτείνουμε κάτι ανάλογο και να στοχεύσουμε τους κλάδους εκτός του ETS. Γιατί συνεχίσει για το ETS, συνεχίζονται, το ETS ενισχύεται, και οπωσδήποτε και βεβαίως και, στον, και υπάρχει και το αποθεματικό της ε, αγοράς και ιδίως στον κλάδο των κτηριών. Τώρα για τους άλλους τομείς αναφερθήκατε στην ε, Ήτρε. Ο κύριος ε, Γκίρεκ ο εισηγητής που ανήκει στη δική σα ομάδα προτείνει έναν στόχο μεταξύ 30 και 40% δεσμευτικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τη σκεφτούμε αυτή την πρόταση. Ίσως έχει μια καλύτερη πιθανότητα να περάσει από την Ολομέλεια. Δεν το ξέρουμε. Πρέπει να δούμε αυτή την συμβιβαστική πρόταση. Ξέρω πως υπάρχουν πολλές ανησυχίες, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι δεν είναι δεσμευτική στο εθνικό επίπεδο η στόχη, που μπορεί να είναι τελικά το αποτέλεσμα της ε, διαδικασίας. Ξέρουμε πως υπάρχουν πολλές ανησυχίες για το πώς θα επιτύχουμε τον συνολικότερο ευρωπαϊκό στόχο. Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε υπό τον όρο η Κομισιόν να συνεχίσει τις προσπάθειες της ε, να αναπτύσσει μηχανισμούς και μέσα για να επιτευχθεί ο στόχος. Και αναφέρομαι ειδικά σε μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και τα μέτρα στον τομέα των μεταφορών. Υπ' αυτόν τον όρο είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτόν τον δεσμευτικό στόχο σε επίπεδο ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συγκίτρια αναφέρθηκε στην σημασία ενεργειακών ελέγχων που πρέπει να ενταθούν. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαστε πεπισμένοι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν τα κατάλληλα μέτρα και κίνητρα. Δηλαδή πρέπει να είναι υποχρεωτικά, δεν είμαστε σίγουροι. Κίνητρα, ναι, οπωσδήποτε. Συμφωνούμε λοιπόν τώρα για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα είναι κάτι το οποίο είναι προσυζήτηση. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, Κυρία εισηγήτρια, συνάδελφοι, έχουμε την πρόταση της εισηγήτρια για το άρθρο 5, το οποίο δεν είναι εντός του πεδίου εφαρμογής που πρότεινε η Κομισιόν. Παρόλα αυτά, ε, είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε ε, με το άρθρο 5 και να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να το διευρύνουμε και να μην το περιορίσουμε, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Οπότε θα σα στηρίξουμε και εκεί. Αυτά, αυτές είναι οι βασικές γραμμές της δικής μας ομάδας. Σα ευχαριστώ, Σα ευχαριστώ κύριε Μπέλετ. Η κυρία Βυσνιεύσκα έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ. κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για την γνωμοδότησή της. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και οι συνεδριάσεις ε, με τους και ηγητές. Φυσικά δεν συμφωνούμε σε όλα. Συμφωνούμε με την αλλαγή του 9α ε, για τις πολυκατοικίες. Ε, θα πρέπει να είναι περιορισμένες οι τεχνικές αλλαγές όταν είναι οικονομικά δυνατές. Μια στιγμή κυρία Βυσνιεύσκα γιατί είχαμε πρόβλημα με τη διερμηνία αρχικά. Μπορείτε να ξαναρχίσετε. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια για το έργο της, για την ομοδότηση και τη συναντήση που οργάνωσε και συμφωνώ με την πρόταση για το άρθρο 9α. Θεωρώ ότι υποχρέωση εφαρμογής ε, τεχνικού εξοπλισμού στις πολυκατοικίες θα πρέπει να είναι περιορισμένος ε, στις ε, περιπτώσεις που από τεχνική άποψη είναι εφικτό και από οικονομική άποψη αποδοτικό. Και φυσικά θα πρέπει να είναι αναλογικό ως προς τα ωφέλη. Οι τεχνικές πτυχές ε, της ενεργειακής απόδοσης είναι διαφοροποιημένες. Εξαρτάται από, τη, από το χρόνο κατασκευής του κτίριου ή της πολυκατοικίας, αλλά και από τη γεωγραφική του θέση πολλές φορές. Οπότε η πολύ αισιόδοξη άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την αλλαγή του τεχνικού εξοπλισμού θα πρέπει να σταθμιστεί με πιο ρεαλιστικά κριτήρια. Επίσης, ε, ε, περιμένω τις προτάσεις ε, της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημείο 5, που δεν περιλαμβάνεται στις τροπολογίες. Υπάρχουν όμως και θέματα που δεν με βρίσκουν σύμφωνα. Αφορά το στόχο του 40% για την ενεργειακή απόδοση ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δεσμευτικό χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τις ε, υποχρεωτικές εθνικές ε, ποσοστώσεις. Βέβαια αυτό συνάδει με προηγούμενε θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν με πλήσει αυτή η πρόταση για τα υποχρεωτικά ποσοστά, αλλά για μένα είναι προβληματικό αυτό το θέμα. Δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι η ενεργειακή απόδοση πραγματικά θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών και θα περιορίσει την εξάρτησή μα στην ενεργειακή. Αλλά πιστεύω παρόλα αυτά ότι στη θέση μα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορου περιορισμού και πολιτικού χαρακτήρα αλλά και τεχνολογικού χαρακτήρα. Από πολιτική άποψη ε, εννοώ τη θέση των κρατών μελών που στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσαν κάποιες πολιτικές κατευθύνσεις με βάση τις συνθήκες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως ξεπερνάει την εντολή που έδωσαν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και είναι αντικείμενο σφοδρή συζήτηση στο Συμβούλιο. Ε, με τόσο υπεραισιόδοξες και υπερφιλόδοξες προτάσεις ε, θα έρθουμε σε διαμάχη με τα κράτη-μέλη. Δεν είμαστε σε θέση να κερδίσουμε σε τέτοια μάχη, κατά τη γνώμη μου. Ε, και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Έχουμε και κάποιους τεχνικούς περιορισμούς και τεχνολογικούς η αποτελεσματικότητα της χρήσης ενέργειας προσκρούσε κάποια όρια ανάλογα με τους τομείς που εξετάζουμε. Και αυτούς τους τεχνικούς περιορισμούς θα πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Για, γι' αυτό και τόσο δραστική αύξηση των ποσοστών δεν με βρίσκει σύμφωνη. Επίσης, ε, το, τροπολογία 21, το, η συνέχεια είναι απαραίτητη. Το άρθρο 7 περιλαμβάνει περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη χρήση του μηχανισμού ελαστικότητας. Γι' αυτό και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί ε, έχετε ανησυχίες έχω προβλήματα με το 21, έχω πρόβλημα και με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο καταπολέμησης της ενεργειακής ένδυας. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά ε, με, είναι η μετακύληση και η επίρρηψη των ευθυνών στα κράτη-μέλη. Μόνο έτσι την καταπολεμάει τη φτώχεια. Και δεν ε, λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι δεν υπάρχει μεθοδολογία για το σωστό υπολογισμό τη κλίμακα του προβλήματο ενεργειακή ένδυα. Φυσικά θα πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις, αλλά δεν μπορούμε να απαιτούμε τέτοιες επενδύσεις από τους πιο απόρους πολίτες. Γιατί οι, επενδύ, οι επενδυτές ε, μετακυλίουν ε, τα, τις ε, ανάγκες τους για την επίτευξη κέρδους σε πιο ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα με το μέτρο που προτείνεται. Αυτά και είμαι ανοιχτή και διαλλακτική στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιάβορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για το σχέδιο κείμενο. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία κατά τη σύνταξη της γνωμοδότησης. Γενικώ συμφωνούμε με το κείμενο. Ε, ακριβώς για, για τον στόχο για τον φιλόδοξο και θεωρούμε ότι τελικά είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Είναι κάτι το οποίο στην πράξη μπορούμε να το πετύχουμε και όχι μόνο από τεχνικής πλευράς. Σήμερα με τη συνθήκη της αγοράς, οπότε αυτός ο πιο φιλοδοξός ε, στόχος αφορά περισσότερη εξοικονομήση ενέργειας. και για τα κρατημέλη γενικώ, αλλά και για τα κτίρια. Να έχουμε αυτούς τους δεσμευτικούς στόχους και θεωρούμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο να φτάσουμε στο να πετύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τα κρατημέλη. Και αυτές οι επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν ούτω ώστε οι ευρωπαϊκές οικονομίες να είναι ανταγωνιστικές και να κάνουν τη διαφορά στα κρατημέλη που έχουν λάβει κάποια τέτοια μέτρα και εκείνοι οι οποίοι υστερούν και έτσι να καλύψουμε την διαφορά που υπάρχει με αυτά τα κρατημέλη. και για τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν καταλαβαίνω γιατί εκείνοι θέλουν να μην υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι, γιατί νομίζω ότι είναι για το δικό τους συμφέρον το να κάνουν ό,τι μπορούν και να έχουμε έτσι πιο φιλόδοξους στόχους και έτσι να έχουμε επενδύσεις για την ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας επίσης, για το άρθρο 7, τα παραθυράκια να κλείσουν, να καλυφθεί και ο τομέας των μεταφορών. Δεν θέλουμε αυτές τις ε, απαλλαγές από το άρθρο 7 και αυτό το όριο του 25% που λέει η συγκίτρια. Αυτό είναι το ελάχιστο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μην εγκριθούν τελικά, να μην περάσουν αυτές οι απαλλαγές. Και όσον αφορά την ε, ενεργειακή φτώχεια, τα κρατημέλη μπορούν να υπολογίζουν ε, στους κοινωτικούς πόρους για το πρόβλημα αυτό. Ναι, έτσι θα πρέπει να αξιοποιούνται οι κοινωτικοί πόροι και να επιδοτούνται κάποια νοικοκυριά μέσω αυτών των πόρων. Τώρα, θα θέλαμε να προσθέσουμε και κάποια άλλα θέματα στην έκθεση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει το ισχύον σύστημα και να υπάρχουν αυτά τα σωρευτικά μέτρα. και επίσης η μακρόπνοη προοπτική επί τη βάση της Συμφωνίας των Παρισίων για το διοξείδιο του άνθρακος και επίσης κάτι άλλο πολύ βασικό είναι η χρηματοδότηση. Από πού προέρχονται τα χρήματα και πώς δαπανούνται όσο αφορά την αποτελεσματική της ενέργειας. Και άρα θα πρέπει να έχουμε χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα σε δύο, τέσσερα χρόνια νομίζω θα έχουν αποδώσει αυτές οι επενδύσεις. Και άρα ε, έτσι θα πρέπει να πείσουμε τον ιδιωτικό τομέα που είναι υπέρ της χρηματοδότησης. Άρα προς τα εκεί να κινηθεί ο ιδιωτικός τομέας και επομένως έτσι να υπάρχει προβλεψιμότητα και σε επίπεδο κρατών μελών. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές διατάξεις και να υποστηριχθούν οι πιο περιθωριοποιημένοι, οι πιο ευάλωτοι και οι Ρωμά. Τέλος δε, νομίζω θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες λύσεις για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις σε κάποια κρατημέλη. Εκεί όπου θα πρέπει τα κίνητρα για αποτελεσματική χρήση της ενέργειας θα πρέπει να διαφοροποιηθούν γιατί υπάρχουν κάποιες παραδόσεις όσον αφορά ε, τα κτίρια, τα μισθωμένα ακίνητα. Και βέβαια θα πρέπει ο οργανισμός να είναι δεσμευτικός, αλλά το βασικό είναι η χρηματοδότηση. Άρα να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους και τους πιο περιθωριοποιημένους από πλευράς εισοδήματος. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω ε, αντί για τον κύριο Πεντιτσίνη. Και να σας πω και τα προσωπικά μου σχόλια όσον αφορά αυτήν την ε, αξιολόγηση της ε, νομοθεσίας για την ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Γενικά, συμφωνούμε με την εισηγήτρια. Συμφωνούμε και με τις ε, τροποποίησεις που έχει επιφέρει όσον αφορά το 40% και τους στόχους. Συμφωνούμε. Θα πρέπει όντως αυτοί οι στόχοι να είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε έτσι υλοποιούμε με συγκεκριμένα μέτρα αυτό το οποίο έχουμε εξαγγείλει ότι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη για να βελτιωθούν όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Οπότε οι καλύτεροι μαθητές, τα κράτη-μέλη που τα πάνε καλύτερα να συνεχίσουν αλλά και οι υπόλοιποι να προσπαθήσουν να πετύχουν τον στόχο που έχουμε τάξει. Ε, βέβαια, η πιο σωστή ενέργεια είναι αυτή που δεν διασπαθίζεται. Και αυτό το διαπιστώνουμε κάθε μέρα, οπότε θα πρέπει να δοθούν τα σχετικά κίνητρα. Ακριβώς αυτό που επανειλημμένα έχει διακηρύξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, συμφωνούμε όσον αφορά το ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποιες ευέλικτες διατάξεις, πρέπει να τις διαγράψουμε, να δούμε τι θα γίνει και με τον τομέα των μεταφορών. Μιλούμε για το 30% κατανάλωσης ενέργεια που αφορά τον τομέα αυτό. Άρα θα πρέπει και ο τομέας αυτός να βοηθήσει όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Απλώς θέλουμε να προσθέσουμε όπως είπαν και οι συνάδελφοι το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Και να προσθέσουμε μόνο το εξής. Εμείς, το κίνημα των πέντε αστέρων, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πετύχουμε να προβλέψουμε για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν οι συνάδελφοι στην Επιτροπή. Τα είπε και ο συνάδελφος Γιάβορ. Και αυτές οι επενδύσεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποδίδουν. Άρα να δοθούν κίνητρα προς τούτο και αυτά τα μέτρα στη, στο σύμφωνο σταθερότητας να καλυφθούν. Και πάλι ευχαριστούμε την εισηγήτρια και ελπίζουμε να συνεχιστεί η καλή συνεργασία μας. Εμείς ευχαριστούμε. Μπόντιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και λαμβάνω τον λόγο. Όχι, αντί της κυρίας Μποντίν που δεν μπορούσε να πραστηλεί κυρία Ντόρνανο. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για τη δουλειά τη. Πρόκειται για ένα σχεδοκειμένο που αφορά την αποτελεσματική χρήση τη ενέργεια, οπότε έτσι τώρα επιβεβαιώνουμε και δίνουμε μια συνέχεια στην οδηγία που ισχύει τώρα και αφορά την ενεργή φτώχεια. Είναι, μέσα στο σωστό δρόμο. Πολλές φορές όμως έχουμε πρόβλημα λόγω των μέτρων λιτότητας που επιβάλλει στους λαούς η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές, η πολιτική μας δεν είναι κατανοητή και δεν ε, ωφελεί από πλευρά σταθερότητα στην ενεργειακή πολιτική. Και αυτό είναι πρόβλημα και για τους επενδυτές και για την βιομηχανία. Όλα αυτά ισχύουν όσον αφορά την ισχύω οδηγία. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσέξει τι θα γίνει όσον αφορά τις ε, ΕΠΑ, όσον αφορά τη Συμφωνία των Παρισίων για την αποτελεσματική ενέργεια. γιατί Τώρα θα υπάρχει ο κίνδυνος να επιταχύνουμε την αποβιομηχάνηση. Επομένως χρειάζεται αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, αλλά αυτό να μην γίνει εις βάρος της βιομηχανίας και εις βάρος της απασχόλησης. Εμείς θα κατεβάσουμε κάποιες τροπολογίες και έτσι αυτή η αναθεώρηση της ε, οδηγίας να καλύψει και αυτά μας τα θέματα. Ή η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Και τώρα, οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Λίζε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Γκούτελαντ με την προετοιμασία. Μπορώ να στήριξω τις αρχικές δηλώσεις να υπενθυμίσω ένα νούμερο. Τα τελευταία χρόνια, κάθε μέρα, δίνουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων. Αν ε, μπορούσαμε να δώσουμε αυτά τα λεφτά στην ε, βιομηχανία μας για να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, ε, θα τα χρησιμοποιούσαμε πολύ καλύτερα. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει διαρροή άνθρακα γιατί επενδύουμε επί τόπου και αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με το ETS, όπου πρέπει να προσέχουμε μην υπάρξει διαρροή άνθρακα. Και θα ήθελα να προσθέσω και για να ανανεώσουμε πηγές ενέργειας, τις οποίες υποστηρίζω, αλλά η εκτίμηση ότι είναι ανεξάντλητες επίσης δεν ισχύει στην περιφερειά μου έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σκεπτικισμός απέναντι στην αιωλική ενέργεια. Οπότε θα επιτύχουμε τους στόχους μας όχι μόνο με ΑΠΕ, αλλά με την μη κατανάλωση ενέργειας. Είναι λοιπόν πολύ καλή η βάση η πρόταση της ε, Κομισιόν και υποστηρίζω κυρίως ε, στο άρθρο 7 να έχουμε μακροπρόθεσμο μακροπρόσμη σιγουριά σχεδιασμού πέρα από το 2020 και 2030. Ότι θέλουμε δηλαδή να στηρίξουμε όσους θα χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα την ενέργεια. Και είναι σημαντικό το ότι έχουμε τώρα την πρόταση του 30% από την Κομισιόν. Γιατί εάν το εφαρμόσουμε όπως προτείνει η Κομισιόν, από αυτό και μόνο έχουμε πληρώσει τους στόχους των Παρισίων, που ήταν στο 27%. Είμαι επιφυλακτικός απέναντι στο 40% ομολογώ ότι το έχει αποφασίσει πολλές φορές το Κοινοβούλιο και την πρώτη φορά το 2014 το είχα υποστηρίξει και εγώ γιατί ήταν τότε επιστημονικά αιτιολογημένο. Έκτοτε όμως έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου και χάθηκαν τρία χρόνια. Και είναι δύσκολο τώρα να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο και δεν θα έχουμε εθνικά δεσμευτικούς στόχους. Ούτως ή άλλως το Συμβούλιο δεν θα ακολουθήσει. Γι' αυτό, όπως είπα, μπέλετε, ένα 35% α, ε, μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Και συμφωνώ Βεβαίω παρά το ότι δεν συμφωνώ με τα υπόλοιπα του κυρίου Γκίρεκ. Τέλος, έχουμε μία ανησυχία στο ΕΛΚ που θα θέλαμε να αναφερθεί. Δεν θέλουμε η πολιτική αυτή να οδηγήσει σε περιορισμό της οικονομικής ανάπτυξης. Δεν μπορεί να λέμε δηλαδή στη βιομηχανία δεν επιτρέπεται να παράγεται ε, λόγω χρήσης ενέργειας. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει τέτοιο. Να μην είναι δηλαδή περιορισμός στην παραγωγή. Τελευταίο, κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή Βιομηχανίας ε, ήδη στις διαπραγματεύσεις ε, μας ε, διαβεβαίωσε πως θα έχουμε ένα άρθρο 53 συν. Βλέπω όμως ότι τώρα το απορρίπτουν. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε και στην ανάγκη να εμπλακεί η διάσκεψη των πρόεδρων. Αυτό αφορά και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και υπήρχε νομίζω και μια σχετική υπόσχεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο Σάικχαουτ. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικός, γιατί με κάλυψε ο συνάδελφος Γιάβορ. Να τονίσω, να τονίσω ότι συνήθως ε, επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, σήμερα, κατά εξαίρεση, θα την επενέσω. Ε, δεν είμαι ακόμη κυβέρνηση. Ξέρω ότι σας σοκάρω, αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την σημασία που έχει αυτή η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της σπουδαιότητας της ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να το λάβουμε απόψη και για την νομοθετική πρόταση. Χαίρομαι που επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαλέγει την αντιπαράθεση με το Συμβούλιο και μένει στη θέση της. Ε, βέβαια, ε, με μισή καρδιά ε, συνεχίζει τον αγώνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι εδώ επανέρχομαι στα, στη συνηθισμένη μου συμπεριφορά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί απέναντι στο Συμβούλιο. Και κοιτάξτε και τον αντίκτυπο επιπτώσεων, αγαπητοί συνάδελφοι, και τι προσφέρει η ενεργειακή απόδοση στην απασχόληση, στην ποιότητα του αέρα, στην ασφάλεια του ενεργειακού ενεφοδιασμού έχουμε τόσους πολλούς δείκτες πέραν της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Πραγματικά είναι πολύ θετική ε, και για όλους επωφελής αυτή η δυνατότητα που μας δίνει η ενεργειακή απόδοση να υλοποιήσουμε τους στόχους του Παρισιού. Και τα λέει ξεκάθαρα η μελέτη επιπτώσεων. Όσο υψηλότερη είναι η στόχη εξοικονόμηση, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Και τα καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε με, τη, με το 40% συντελεστή ε, ποσοστό ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σα ευχαριστούμε που πιέσετε το Συμβούλιο. Εμεί είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι γιατί συμφωνούμε με τη μελέτη επιπτώσεων και θέλουμε η δεσμευτικότητα να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο, γιατί παρά ε, έχει εμπιστοσύνη στη, στα κράτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ε, προτιμούμε και σε εθνικό επίπεδο να είναι υποχρεωτική δεσμευτική στόχη. Και μετά από τέτοια θετικότητα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένω κάποια ανταλλάγματα. Και αυτά αφορούν τις μεταφορές συμφωνώ με την πρόταση Ηγήτριας να συμπεριλάβουμε και τις μεταφορές, γιατί εκεί είναι που χάνουμε σε απόδοση ενεργειακή. Και φυσικά να συμπληρώσουμε αυτή την πρόταση με, ενεργη... με προτάσεις πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε και ο τομέας των μεταφορών με συγκεκριμένους στόχους να συμβάλλουν και οι μεταφορές στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Θέλουμε λοιπόν φιλόδοξους στόχους όπως αυτούς που έχουμε είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιου στόχου και για το 2025. Όσο πιο νωρίς συμπεριλάβουμε τι μεταφορέ, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. Και πραγματικά ε, εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση. Μετά λοιπόν τα θετικά μου σχόλια προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένω και κάποια ανταλλάγματα ε, για να μην ε, ξενήσω τόσο πολύ του συναδέλφου με τόσο διαφορετική στάση. Ο κύριο Φλόρεντ. Φοβερή αυτή η σύνδεση κομισιών και έτσι η Ολλανδική αυτή σύνδεση. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, γιατί έχουμε επιβάλει υψηλούς στόχους στην βιομηχανία και δεν είμαστε πολύ ενεργοί σε αυτόν τον τομέα. Τώρα για το 40% δεν είναι αυτό το αποφασιστικό. Αποφασιστικό είναι να διαπιστώσουμε ότι στην χώρα μου, την Αυστρία και στην Ολλανδία επί σειρά ετών προσπαθούμε να επιτύχουμε το θέμα αυτό στα κτίρια και αποτυγχάνουμε. Στη χώρα μου υπάρχουν χρήματα ναι. κάτω από 1%, κάτω από 0% επιτόκιο και δεν ε, γίνονται οι επενδύσεις. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα ε, αντίληψης και συνείδησης. Δηλαδή αν ε, δεν έχουμε πιστεί εδώ μέσα, φανταστείτε τι γίνεται έξω από αυτήν την εύσοα. Οπότε δεν ξέρω εάν θα γίνει ε, κάτι τέτοιο υποχρεωτικό αν δεν καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε να κάνει ο κόσμος κάτι μόνος του. Δηλαδή όταν, υπάρχουν τόσο, όταν υπάρχει τόσο φτηνή χρηματοδότηση και δεν το κάνει ο κόσμος, το πρόβλημα δεν είναι η γραφειοκρατία, είναι ότι δεν πείσαμε τον κόσμο. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμένα. Σας ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι των Παρισίων θα παίξει σημαντικό ρόλο η ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Η αρχική στόχη ε, κατά 20% βελτίωση ε, δεν επαρκούν πλέον, ειδικά εφόσον έφυγε ο Τραμπ από τους στόχους. Ε, είναι ακόμη σημαντικότερο η Ευρώπη να είναι φιλόδοξη. Γι' αυτό πρέπει να αυξηθεί η ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Εντάξει, 40% μπορεί να μην το επιτύχουμε, πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, να δούμε τι θα γίνει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, σωστά. Ε, γι' αυτό όμως χρειαζόμαστε χάλιβα. Ο χάλιβας όμως απαιτεί ενέργεια. Δηλαδή πρέπει να παραχθεί κάπως και ο χάλιβας. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να είμαστε κάπως ισορροπημένοι, να πούμε ναι, θέμε φιλοδοξία, ναι, ψηλότερους στόχους, αλλά πρέπει να έχουμε και ευελιξία και κάποιο περιθώριο για την ε, βιομηχανία. Οι μεταφορές πράγματι σημαντικές ε, για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Υπάρχει νομίζω η απομάκρυνση στον κλάδο αυτόν από τον άνθρακα. Ε, εντάξει υπάρχουν πολλά πρέπει να γίνουν, σωστά, αλλά πρέπει να δούμε το σύνολο γιατί ε, οι μεταφορές ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουν και λιγότερη ενέργεια αλλά να έχουν και εξυπνότερα συστήματα μεταφορών νέα υλικά ε, ενιαίος ευρωπαϊκός εναέριος χώρος διάφορα πράγματα. Και ε, πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε ε, όχι μόνο να ε, βλέπουμε το θέμα από την σκοπιά του περιβάλλοντος, αλλά το τι μπορούμε να προσφέρουμε στην βιομηχανία και να ενημερώσουμε τον, τον κόσμο. Συμφωνεί ο Μπασάικ Χάουτ, ενδιαφέρον αυτό. Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Θα καταθέσω και κάποιε τροπολογίε, αλλά ευχαριστώ ήδη την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια. Ε, υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τους δεσμευτικούς στόχους. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πρόσφατη μελέτη της Κομισιόν από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο που δείχνει ότι ο στόχος του 20% του 2020 είχε επιτευχθεί ήδη το 2014 και θεωρώ ότι αυτό είναι επιχείρημα για μεγαλύτερη φιλοδοξία για το 2030 και πρέπει να ενισχύσει την αποφασιστικότητά μας για ένα στόχο 40%. Κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αφορά το πώς θα εξελίψουμε τα παραθυράκια και τις ευελιξίες. Ειδικά δεδομένου του ότι το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις ε, έκανε, ε, εξασθένησε κατά πολύ την θέση μας μέσω διαφόρων εξαιρέσεων που πρέπει να φύγουν από τη νέα οδηγία. Ειδικά καθώς η μελέτη του EPRS έδειξε ότι στην πραγματικότητα τα και αυτά οδήγησαν στο να επιτευχθεί μόνο ο μισός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας. Για την ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων θεωρώ ότι πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα ο δημόσιος τομέας και εδώ πέρα συμφωνώ με την εισηγήτρια όταν λέει ότι θα πρέπει να τεθεί ο στόχος του 3% των δημοσίων κτηρίων που θα πρέπει να ανακαινίζονται κάθε χρόνο σε όλα τα δημόσια κτίρια, όχι μόνο τα κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης και πρέπει να φροντίσουμε ο εισηγητής να είναι παρόν και κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και του τριμερούς διαλόγου. Ευχαριστώ και πάλι. Μάλιστα, ναι, δεν έχουμε κάποια απάντηση από την Ήτρε. Για το άρθρο 53 συν, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Ο κ. Πολ Χάτσον τώρα από την Επιτροπή για να αντιδράσει τα όσα ακούστηκαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα σας. Με πολλά συμφωνώ. Δεν θα παταλήσω τον χρόνο σας. Συμφωνούμε με τα όσα ακούστηκαν για τα ωφέλη της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ειδικά όσον αφορά τα αερία του θερμοκηπίου. Επίσης ε, συμφωνούμε με αρκετούς ευρωβουλευτέ ε, για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλόρενς. Ε, πρέπει να υπάρχει εφαρμογή. Δεν αρκούν οι φιλόδοξοι στόχοι και άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε με ε, τον κόσμο και όχι να επιβάλλουμε πράγματα. Τώρα, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα, δεν θα αναφερθώ στα επίπεδα των στόχων, τα δεσμευτικό χαρακτήρα κτλ. Κάποια από αυτά είναι κάπως επίμαχα ακόμα. Θα συμφωνήσω όμως με τον κύριο Μπέλετ ότι η εθνική δεσμευτική στόχη είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δεν μας χρειάζεται εδώ πέρα. Έχουμε άλλα εργαλεία, ανανεώσιμη ενέργεια όπως αυτά τα οποία αναφέρατε, οικολογικός σχεδιασμός, ε, cars κτλ και μπορούμε βεβαίω να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δράση. Και βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να προχωρήσουν παραπέρα. Δεν προτείνουμε λοιπόν δεσμευτικού στόχου, δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Για την ενεργειακή φτώχεια, για να απαντήσω στην κυρία Βυσνιεύσκα, οπωσδήποτε δεν λέμε ότι η ε, νομοθεσία η σχετική πρέπει να αντικαταστήσει τι εθνικέ κοινωνικέ πολιτικέ για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζει το κάθε κράτο μέλο με το δικό του τρόπο. Ε, δεν είναι θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ένα μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα είναι να μην σπαταλάνε τα άτομα με χαμηλό εισόδημα λεφτά για ενέργεια η οποία σπαταλάται γιατί δεν υπάρχει η σωστή μόνωση. Είτε νοικιάζουν είτε είναι δικό τους το σπίτι. χωρίς να είναι βεβαίω αυτή η πηγή τη ενεργειακή ένδυας. Αλλά σε ένα πακέτο απελευθέρωσης των τιμών τη ενέργεια, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δώσουμε και εκεί πέρα κάποιο βάρο. Συμφωνούμε με τον κύριο Γιάβορ για την σημασία της χρηματοδότησης. Κάνουμε πολλά πράγματα εκτός αυτής της ε, πρότασης για να μειωθεί η αίσθηση του κινδύνου στους επενδυτές ε, να προσπαθήσουμε να διασπείρουμε τον κίνδυνο και θα πρέπει ακριβώς να δώσουμε βάρος στην ιδιωτική χρηματοδότηση και το πώς θα την προσελκύσουμε αντί να δίνουμε κατευθείαν επιχορηγήσεις. Δεν συμφωνούμε με την κυρία Ήβη ότι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να μετράει για το σύμφωνο ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει να γίνεται ε, διακριτική μεταχείριση, αλλά ούτε και να εξαιρεθεί. Ε, Κύριο Σάικχαουτ, τι χαρά, τι χαρά να μας επενείτε εσείς. Ε, πραγματικά θα το γράψω πρώτο-πρώτο στην έκθεσή μου. Για το θέμα των μεταφορών όμως υπάρχουν και άλλες δήματα πέρα από αυτήν την πρόταση και μάλιστα θα ζητήσουμε ακριβώς να στηριχθούν οι προτάσεις που έχουμε κάνει για να προωθηθεί η σχετική κινητικότητα και όπου ακριβώς έχουμε το πρόβλημα για να γίνει το επόμενο βήμα. Θέλω να πω επίσης πως χαιρόμαστε για αυτό το οποίο μας είπε ο κ. άλλοι για την μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Συμφωνούμε να έχουμε μια προοπτική και μέρα από το 2030 και ελπίζω πράγματι το κοινοβούλιο να μας στηρίξει εδώ. Τέλος, δύο τεχνικά ζητήματα που πρέπει να πω. Υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο ενεργειακής νομοθεσία και η Κομισιόν ζητάει και από τους δύο συνομοθέτες να παραμείνουμε εντός του πεδίου που προτείνει η Κομισιόν. Οπότε δεν στηρίζουμε την πρόταση της εισηγήτριας ε, στην τροπολογία 17 να δούμε το άρθρο 5, δηλαδή να πάμε από τα κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης σε όλα τα δημόσια κτίρια. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποια ουσία, αλλά τελικά θα δημιουργήσει και άλλες συζητήσεις που δεν χρειάζονται τώρα για το άρθρο 8 για τους ενεργειακούς ελέγχους. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε την ουσία των τροπολογιών 29 με 31, αλλά δεν θεωρούμε ότι δικαιολογούνται τώρα νέε συζητήσει. Και για το άρθρο 8, πείσαμε το Συμβούλιο σε παρόμοιες καταστάσεις να μην ξανανοίξει το διατακτικό, αλλά να συνεργαστεί μαζί μας σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκούτλαντ, η συγγετριά μας για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους ως προς την γνωμοδότηση. Δεν πρόκειται να απαντήσω σε όλα τα σχόλια τα επιμέρους, αλλά χαίρομαι που σε πολλά σημεία συμφωνούμε. Θα πω λίγα λόγια για τους δεσμευτικούς στόχους και τη φιλοδοξία. Πρέπει να είναι σημαντικό τμήμα της έκθεσης αυτή η φιλόδοξη στόχη. Αυτό που παρατήρησα και εγώ προσωπικά είναι ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι θα προτιμούσαν μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα στην αγορά. Αυτή την εντύπωση αποκόμισα από τις ε, πολλές συναντήσεις που είχαμε ενδιαφερόμενους και το μήνυμα της εξασφάλισης επαρκούς επένδυσης ε, σε νέες τεχνολογίες και νέες λύσεις ε, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ήταν το μήνυμα που έλαβανα παντού. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το εξασφαλίσουμε με δεσμευτικούς στόχους, αυτή την προβλεψιμότητα και την σαφήνεια. Και έτσι θα εξασφαλίσουμε και συμμόρφωση των κρατών μελών με τα ευρωπαϊκά μέτρα. Γι' αυτό είμαι υπέρ των δεσμευτικών στόχων και σε εθνικό επίπεδο. Ως προς το επίπεδο φιλοδοξίας, θεωρώ ότι η ενεργειακή απόδοση είναι από τους πιο σημαντικούς και όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τους πιο χρήσιμους ε, μηχανισμούς ε, που έχουμε, όχι μόνο για να υλοποιήσουμε τη Συμφωνία του Παρισιού, αλλά είναι και ο κλάδος που θα μας εξασφαλίσει τα πιο θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και θα συμβάλλει ανάλογα με το επίπεδο των φιλοδοξιών μας στην εξασφάλιση περισσότερων θέσεων απασχόλησης, μεγαλύτερης ασφάλειας και καλύτερης υγείας ε, των συμπολιτών. Ε, ε, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση έχουμε 2,5 με τέσσερις φορές περισσότερη αύξηση των θέσεων απασχόλησης σχέση με άλλους κλάδους. Και ξέρουμε πόσο απεγνωσμένοι είναι οι Ευρωπαίοι άνεργοι και πόσο λαχταρούν να έχουν μια δουλειά. Γι' αυτό και θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπαθίες μας. Επίσης, ε, με την πρόταση για την ενεργειακή απόδοση θα μειώσουμε αισθητά τι ε, εισαγωγέ ενεργειακών προϊόντων. Ε, για την περίοδο 2021 με 2030 η μείωση στι εισαγωγέ ορυκτών καυσίμων θα μα εξοικονομήσει 2,88 δισεκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντα και πάλι στην ενεργειακή μας ασφάλεια. Και τέλος, πολύ σημαντικό όμω θέμα και πολλαπλασιάζεται τα ωφέλη το πιο χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό παράδειγμα για τα ωφέλη της ενεργειακής απόδοσης ε, αφορούν την υγεία. Το προσδόκιμο ζωής, χάρη στην πρόταση της ενεργειακής ε, απόδοσης, θα αυξηθεί και θα, θα εξοικονομήσουμε 17 δισεκατομμύρια από τι δαπάνε υγείας χάρη στη βελτίωση της, ατμοσφαιρικής του, της ποιότητας του αέρα. Θέλω λοιπόν να είμαστε συνεπείς και να τιμήσουμε τις ε, ηλιμένες αποφάσεις, οι πρόσφατες αποφάσεις ήταν του περασμένου έτους και να επιμείνουμε σε αυτό το φιλόδοξο στόχο του 40% για την ενεργειακή απόδοση. Καταλαβαίνω τα σχόλιά σας για τις αντιθέσεις ε, του Συμβουλίου, αλλά αυτό το, το χαρακτήρα έχουν οι διαπραγματεύσεις. Αν από την αρχή νερώσουμε το κρασί μας και έχουμε ε, χαμηλότερες φιλοδοξίες, την πορεία των διαπραγματεύσεων θα χρειαστεί να τις ε, περικόψουμε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε από την αρχή υψηλέ ε, φιλοδοξίες για να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Δεν συμφωνώ ότι εμείς θα πρέπει να μειώσουμε από την αρχή του τριμερούς διαλόγου τις φιλοδοξίες μας. Έτσι αποδυναμώνουμε τη διαπραγματευτική μας ισχύ. Ευχαριστώ. Πολύ συγκινητικές αυτές οι δηλώσεις και αποφασιστικές επίσης. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Να μην ξεχνάμε την προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. 14 Ιουνίου, 11 το μεσημέρι. Και 7 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Είστε έτοιμοι να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχετε τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες. Το πρώτο σημείο είναι η ψηφοφορία για την εντολή για το διμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Η δεύτερη ψηφοφορία αφορά την έκθεση Γιάβορ για την εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη σε σχέση με την πρόληψη και τη διόρθωση της περιβαλλοντικής ζημίας. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 6 παρακαλώ. Τέλος, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική παριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 5. Υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την προφορική τροπολογία. Θέλετε να τη διαβάσετε. Την γνωρίζετε. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Μήπως όχι, οπότε ψηφίζουμε τη συμβαστική με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 35. Άρχεται ψυχοφορία ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ομολογώ δεν κατάλαβα πώς ψηφίζουν οι σοσιαλιστές, αλλά αυτό είδα. θέλω ψηφοφορία. Απορρίπτεται, αλλά ήταν ισοπαλία. Ε, ισοπαλία υπέρ και κατά. Τροπολογία 37. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα για την 52. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 50, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Γιάβορ. Και ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες μας. So, dear colleagues, Κύριος Γιάβορ, συνεχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ. Όποιος δεν ε, θα συμμετάσχει σε αυτό το σημείο τη να, να αποχωρήσει. Και το επόμενο σημείο της διάταξη είναι τα νομοθετικά μέτρα, ώστε να υπάρξει προστασία των καταγγελόντων για το δημόσιο συμφέρον και ο εισηγητής κ. Φλάνεγκαν έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου ικανοποίηση ανέλαβα αυτή την ε, έκθεση και όλοι να ασχοληθεί με τους καταγγέλλοντες μου λένε ότι είναι κάποιοι θαραλέοι ε, και θα πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να τους προστατεύσουμε και θεωρητικά δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα προς τούτο. Επίσης όλοι θα σας πούν ότι όντως πρόκειται για κάποιους που έχουν το κουράγιο αλλά δεν θα έπρεπε να απαιτείται κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να θεωρείται φυσιολογικό στα πλαίσια της δουλειάς κάποιου που όταν διαπιστώσει ότι κάτι πάει στραβά να το καταγγέλουν. Αλλά ο λόγος το ότι χρειάζονται ιδιαίτερο θάρρος είναι ότι κάποιος οφείλει να τους προστατεύσει. Ε, αν όμως υπήρχε κάτι τέτοιο ε, δεν θα χρειάζεται να κάνουμε αυτή την έκθεση τέλος πάντων. Οπότε δεν υπάρχει τώρα επαρκής προστασία και αυτό οδηγεί στο ότι δεν έχουμε ε, για το περιβάλλον, για τη διατροφική ασφάλεια, για την υγεία, ε, ε, ικανοποιητική εφαρμογή της νομοθεσίας μας. Επομένως θεωρούμε ότι αν προστατεύσουμε τους καταγγέλλοντες θα έχουμε καλύτερη υλοποίηση των σχετικών πολιτικών. Επίσης λέω ότι χρειάζεται σωστή νομοθεσία και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και λέμε ότι ε, κάποια κράτη-μέλη δεν κάνουν ε, αυτό το οποίο χρειάζεται και ενώ θα έπρεπε να εξασφαλίσουν προστασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνω Επιτροπή να υποβάλει κάποια πρόταση οδηγίες για την προστασία αυτών. Ε, στο έκτο σημείο λέμε ότι υπογραμμίζουν τα επιβαλλοντικά εγκλήματα για δημόσια υγεία, γεννήτρο φήμων. θα πρέπει να εμπίπτουν σε αυτά τα μέσα. Στο έβδομο σημείο λέμε ότι η νομοθεσία για την προστασία των καταγγελώντων, θα πρέπει να είναι άμεση για τους αδέλφους, συγγενείς τους, για κάθε ενέργεια και κάθε αντίπεινα. Επί στο 8 λέμε ότι ο ορισμός του καταγγέλους δεν θα πρέπει να είναι στενός, να μην αφορά μόνο ορισμένους τομείς και θα πρέπει επίσης να έχουν ίση προστασία σε και τομέα ίση ίση προστασία και στους τομείς. Στο δένατο σημείο λέμε ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφή διαδικασία για κάθε ε, χειρισμό των αναφερομένων πληροφοριών. Οπότε τα πράγματα είναι προφανή συμπερασματικά. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να προβλεφθεί και νομίζουμε ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση προς τούτο τότε ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Σας ευχαριστούμε και τώρα για τις πολιτικές ομάδες. Πρώτα το ΕΛΚ. Τουρκάνου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η έκθεση που αφορά τους καταγγέλλοντες εγκρίθηκε στην ε, Νομική Επιτροπή το Σεπτέμβριο. Φέτος έχουμε εισηγεί την κυρία Ροζιέρ και είπαμε ότι πρόκειται για θέμα προτεραιότητας για μας. Μια που το θέμα αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, τον πλουραλισμό των απόψεων είναι σημαντικό για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει να πετύχουμε την ε, ε, κατάλληλη ισορροπία γιατί οι καταγγέλλοντες βοηθούν πάρα πολύ την πολιτική προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της διατροφικής ασφάλειας. Η προστασία των καταγγελόντων θα οδηγήσει σε περισσότερη διατροφική ασφάλεια. Τώρα, έχω κάποιες τροπολογίες και θα συνεργαστούμε με όλους όσους ασχολούνται με το θέμα. Σε ευχαριστώ. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η κυρία Τζέντας. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο από την Ιρλανδία για το σχέδιο γνωμοδότησης. Είμαστε και οι δύο από μια χώρα όπου τα αντίπεινα κατά των καταγγελόντων ήταν ρουτίνα. Και οπωσδήποτε έχουμε επηρεαστεί από το πώς έχει επηρεάσει αυτό την εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας. Είναι δύσκολο βεβαίως να μετρηθεί κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι ε, αυτό μας κόστισε μία από τις πιο μεγάλες τραπεζικές κρίσεις στην πρόσφατη ιστορία, η οποία οδήγησε σε λιτότητα, αλλά ακόμα και σε μία κρίση πνευματικής υγείας και αυτοκτονιών. Και ταυτόχρονα βεβαίως είχαμε και μια προσπάθεια να σπηλωθεί η τιμή της κοινωνικής λειτουργού η οποία ε, το αποκάλυψε. Το ίδιο και με την υπόθεση του αλογίσιου κρέατος. Λοιπόν, η νομοθεσία αυτή ε, ξεκίνησε να ισχύει το 2013, αλλά ο νόμος από μόνος του δεν επαρκεί για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των καταγγελόντων, ειδικά όταν έχουμε κάποιες αποκτηνωμένες ε, θεσμικές κουλτούρες. Γι' αυτό τη κράτη-μέλη έχουν νομοθετήσει σε μεγάλο βαθμό κάποια νομική προστασία, κάτι το οποίο βεβαίως οδηγεί σε έναν κατακαιρματισμό του νομικού τοπίου. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε διαφορετικές αντιμετωπίσεις ε, σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, δημόσιας ε, υγείας και ασφάλειας των τροφίμων αναλόγως με την προστασία που απολαμβάνει ο καθένας. Γι' αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε με τον συνάδελφο εδώ πέρα η Κομισιόν να προτείνει μια οριζόντια οδηγία για το θέμα αυτό. Όλοι είδαμε το θέαμα της δίκης του LuxLeaks όπου κάθισαν στο σκαμνί οι καταγγέλλοντες επειδή παραβίασαν τους νόμους εμπιστευτικότητας του Λουξεμβούργου σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καταδικάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ο κύριος Γιούνκερ έγινε πρόεδρος της Κομισιόν και η PwC έχει κερδίσει συμβόλαια εκατομμυρίων με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εγώ προσωπικά απέριψα την οδηγία περί εμπορικών μυστικών και την απέριψα γιατί αυτά τα οποία προέβλεπε για την προστασία των καταγγελόντων που δρούν καλή την πίστη, αλλά και όσων στα μήμια αποκαλύπτουν αυτά τα ζητήματα ήταν ανεπαρκήσαν και οφείλω να επενέσω την δουλειά των συναδέλφων και των σοσιαλιστών συναδέλφων και του κυρίου Κοφεράτη, αλλά επίσης ήταν κακός ιονός το ότι απαλλάξαμε την Κομισιόν και έτσι στείλαμε ένα ανησυχητικό μήνυμα σε καταγγέλλοντες στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραπέρα. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανεπάρκεια και άλλες, θα πρέπει να πιέσουμε την Κομισιό να προτείνει μια οδηγία η οποία θα προβλέπει έναν ευρύτερο ορισμό της ε, καταγγελίας σε διάφορους κλάδους με νομική βεβαιότητα σε ολόκληρη την Ένωση. Η περιπλοκότητα βεβαίως ε, του ζητήματος ε, δεν εμπόδισε την Κομισιόν να νομοθετήσει για τα εμπορικά μυστικά. Γιατί την εμποδίζει εδώ. Έχει περάσει λοιπόν, ε, πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί αυτή η ασυμμέτρια που, τι λέει, η ασυμμετρία με που υπάρχει στον τομέα αυτόν και θα συνεργαστώ με τους ε, σκιώδεις συγητές. Σας ευχαριστώ. Δεν... Ε, σκιώδεις συγητές από το ECR και τις άλλες ομάδες. Οπότε ε, θα μιλήσω εγώ από τους πράσινους. Υπάρχει κάτι το σημαντικό αυτό δεν είναι μια ηθική υποχρέωση ή κάτι το καλό, αλλά τελικά προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους καταγγελτές γιατί δρούν ε, εξ του κοινού και προστατεύουν εμάς ως κοινό, ως κοινωνία και θεωρώ ότι τελικά πρέπει να αποδείξουμε ότι οι καταγγέλλοντες που ρισκάρουν πολλά πράγματα Ε, μπορούν να βασίζονται σε εμάς. Είμαστε στο πλευρό τους και όχι στο πλευρό όσων διαπράττουν αδικήματα. Από αυτή την ε, σκοπιά οφείλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φλάναγκαν για την εξαιρετική έκθεση και θα ήθελα να τονίσω κάποια ε, σημεία με τα οποία συμφωνώ. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας στην Ένωση και βεβαίως υπάρχει διαφορετικό επίπεδο νομοθεσίας. Και οι περιπτώσεις ε, τις οποίες αναφέρουν οι καταγγέλλοντες συχνά έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και δεν μπορούν να είναι σίγουροι ποια νομοθεσία θα ισχύσει. Επίσης είναι σημαντικό να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Εγώ θα τα προσθέσω με τροπολογίες. Θα τονίσω την ε, διασυνοριακή φύση ακριβώς ε, του πράγματος, γιατί η φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων συχνά δεν περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος, οπότε ούτε και οι καταγγελίες. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι φυστάμενες διατάξεις στο επίπεδο των κρατών μελών ε, έχουν περιορισμένο εύρος, καλύπτουν κάποιους κλάδους και περιπτώσεις και αφήνουν έτσι παραθυράκια και οδηγούν σε νομική αβεβαιότητα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μεγάλη σημασία έχει ακριβώ το να προλάβουμε εγκαίρως Κάποιου ε, περιβαλλοντικούς κινδύνους, όχι μόνο να τιμωρήσουμε όσου ρηπαίνουν, αλλά να προλάβουμε τη ζημιά του περιβάλλοντος. Ε, και αυτό θα γίνει αν προστατεύονται και ενθαρρύνονται οι καταγγέλλοντε. Και τέλος, να πω, και το αναφέρθηκε και από την κυρία Τσίλντερς αυτό, σχετική οδηγία. Η Επιτροπή Προπολογισμού ασχολείται με αυτή την έκθεση, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αλλά η κλαδική νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει πάλι ένα μοσαϊκό ε, νομοθεσίας σε διαφορετικούς τομείς. Και οπότε θα μεταφέρουμε αυτό το οποίο έχουμε τώρα στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν μια οριζόντια οδηγία που θα έχει κάποιες ε, σοβαρές ελάχιστες απαιτήσει για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την ε, συνεργασία με την... Ε, τον εισηγητή για τις περιβαλλοντικές πτυχές των καταγγελιών. Σας ευχαριστώ. Ξαναγίνομαι τώρα πρόεδρος και δίνω το λόγο στην κυρία Τανανό, την σκιώδη του ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Φλάναγκαν, για την παρουσίαση και φυσικά προσυπογράφω τη γνωμοδότησή σας γιατί οι καταγγέλλοντες έχουν αποκαλύψει και περιβαλλοντικά σκάδαλα και σκάδαλα στην υγεία ε, τοξικότητα κάποιων ουσιών και βαρέων μετάλλων. Επίσης, στρέφονται κατά τα κατά των ιδιωτικών συμφερόντων και μερικές φορές οι συνέπειες και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο είναι πολύ δυσάρεστος. Γι' αυτό θέλω να αναλάβουμε κάποιες ε, γενναίες ε, δράσεις και να προστατεύσουμε τέτοιες θαραλές συμπεριφοράς. Τα άρθρα 1-5 της οδηγίας για το εμπορικό απόρριτο περιέλαβαν κάποιες μνήες που αφορούν και τους καταγγέλλοντες στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Λοιπόν, έχουμε και ε, συγκεκριμένη αναφορά, αλλά δεν αρκεί οδηγία αυτή για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας για τους καταγγέλλοντες. Είμαι λοιπόν υπέρ της ιδέας της θέσπισης ε, κατάλληλων νομικών ε, μέσων που θα προστατεύουν καλύτερα τους καταγγέλλοντος. Θα καταθέσω και τροπολογίες στην ε, στο σχέδιο γνωμοδότης, γιατί θα πρέπει να επιμείνουμε στην προστασία της ανωνυμίας των καταγγελόντων, ώστε να αποφύγουμε διώξεις βάρος τους. Επίσης, θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να εξασφαλίσουμε το, την απόρριτη επεξεργασία των καταγγελιών. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταγγελόντων από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα ή τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, γιατί έχουν επισημάνει συγκρούσεις συμφερόντων ε, για επιστημονικό προσωπικό της, ε, του Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων. Επίσης, θα πρέπει να εξαιρέσουμε από το πίδιο εφαρμογής οδηγίας κάποιες ε, εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την προάσπιση των ζωτικών συμφερόντων των κρατών μελών. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να παρακινούνται να δημοσιεύουν τέτοιου είδους πληροφορίες που αφορούν ζωτικά εθνικά συμφέροντα, γιατί κάτι τέτοιο δεν συνάδει με το δημόσιο συμφέρον. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σούλαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ενημερώσω για την πορεία του θέματος αυτού. Όπως ξέρετε παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς αυτό το θέμα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, παρακολουθώντας και το σχέδιο εργασιών του 2017. Ε, εξετάζουμε το κατά πόσο είναι εφικτές νέες δράσεις και ποια θα είναι η νομική τους εμβέλεια είτε μέσω πολιτικών, ίσω κάποιων οριζόντιων ή τομεακών νομοθετικών δράσεων για να ενισχύσουμε την προστασία των καταγγελόντων. Φυσικά, με πλήρη σεβασμό τη αρχή της επικουρικότητα. Με βάση λοιπόν αυτό το σκοπό έχουμε ξεκινήσει δημόσιε διαβουλεύσεις 3 Μαρτίου που ολοκληρώθηκαν στι 29 Μαου και τη ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης εκπονούμε μελέτη για τη συγκέντρωση εμπειρικών στοιχείων σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που έχουν μέτρα προστασίας ε, καταγγελόντων ε, για την ανείχνευση ατασταλιών για δικοπραξιών. Χάρη σε όλες αυτές τις πληροφορίες ε, θα καταλήξουμε σε περιστατωμένη άποψη για το τι πολιτικές και μέτρα ενδεχομένω και νομοθετικά απαιτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελπίζω ήδη από τον Ιούλιο να έχουμε τα αποτελέσματα και της δημόσιας διαβούλευσης και της μελέτης οπότε να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των πορισμάτων. Ευχαριστώ. Επαναρχόμαστε στον εισηγητή μας και πάλι τον κύριο Φλάναγκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για τις πληροφορίες που μας έδωσαν και τα σχόλια. Εγώ δεν είχα πολλές επαφές με καταγγέλλοντες. Φαντάζομαι ότι εσείς είχατε περισσότερες εμπειρίες. Πάντως, ε, ε, όταν ε, έχω επαφή μαζί τους, ε, εξετάζω αν τα ψυχικά προβλήματα προηγούνται της αποκάλυψης του σκανδάλου ή έπονται. Πάντως, πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι υφίστανται ψυχική καταπίεση από αυτούς που έχουν καταγγείλει. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η παρενόχληση πραγματική και ψυχική. Και είχα πολλές επαφές στην Ιρλανδία που χρειάστηκε να έρχονται με αλεξίσφαιρα στο γραφείο μου. Εγώ τους ε, έλεγα όταν μου ζητούσαν συμβουλές, κρατήστε το σώμα σας κλειστό. Μην ε, είστε χαζοί, θα καταστρέψετε τη ζωή σας. Και σας το λέω γιατί ε, μέχρι και συκοφαντίες για παιδεραστία είχαν γίνει βάρο βάρος καταγγελόντων. Μάλιστα, επειδή δεν είχαμε babysitter, έφερα την 11χρονη κόρη μου σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή στην Ιρλανδία, όπου ένας καταγγέλων ε, μιλούσε για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και μετά την ακρόαση ακόμη και η κόρη μου 11 χρονών κατάλαβε να σε πρόκειται. Μου είπε «Μπαμπάκα, ο άνθρωπος αυτός ε, έχασε τη δουλειά του στην τράπεζα γιατί αν δούλευε σε άλλη τράπεζα και έκανε η τράπεζα κάτι κακό θα έλεγε την αλήθεια και θα τους ε, δημιουργούσε προβλήματα. Ναι, είπα κοριτσάκι μου, έχεις δίκιο. Αν και ενα εντεκάχρονο παιδί είναι στη θέση να καταλάβει τις δυνάμεις που κινούνται όταν ε, ένας καταγγέλων κάνει μια καταγγελία, εμείς Πώς είναι δυνατόν να εθελοτυφλούμε, γιατί αυτό φαίνεται να γίνεται από πολλούς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι και η ώρα να αναλάβουμε επιτέλους δράση για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Και εντάξει, μιλούμε για τους καταγγέλλοντες στον τομέα της υγείας ή σε άλλους κλάδους, αλλά θα πρέπει να καλύψουμε όλους τους κλάδους ε, όταν συζητάμε αυτό το θέμα, γιατί ε, έχει, έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία όλων, ό,τι αντικείμενο και να έχουν οι καταγγελίες, στο περιβάλλον, την υγεία, την ε, γεωργία, το χρηματοοικονομικό τομέα. Σίγουρα επηρεάζεται αρνητικά η υγεία των καταγγελόντων, ό,τι χαρακτήρα και να έχει η καταγγελία τους. Ευχαριστώ. Η προθεσμία για την καταβολή τροπολογιών, για την κατάσταση τροπολογιών είναι 16 Ιουνίου, 11 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 11 Ιουλίου και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στις 28 Σεπτεμβρίου. Αναμένουμε ε, να ψηφιστεί η έκθεση στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου, στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με την οδηγία για τα πτηνά και τα διαιτήματα και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η προτινόμενη διαδικασία για την ανταλλαγή απόψεων είναι προβλέπει πρώτα παρουσίαση του κυρίου Ρώσα από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Είναι διευθυντής ε, τη, της τέταρτης διεύθυνσης για το φυσικό κεφάλαιο, κύριος Δελγάντο Ρώσα. Μετά την παρουσίαση του κύριου Ρώσα θα γίνει συζήτηση με τους παρόντες φυσικά. Ο κύριος Ρώσα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Μας δίνει την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσουμε αυτό το πρόγραμμα δράσης και να το συζητήσουμε όσον αφορά την φύση και την οικονομία Οπότε να σας παρουσιάσω αυτό το πρόγραμμα. Όπως ξέρετε έχουμε ε, αυτά τα δελτία, δημοσι... τα έχουμε δημοσιεύσει. Και το πώς οι βουλευτές έχουν διαφερθεί δείχνει τη σημασία του θέματος. Οι στόχοι επομένως του προγράμματος ε, πηγάζουν από τον έλεγχο των ισχυουσών οδηγιών. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή τους. Θα γίνει με τα και να δούμε και πώς συμβάλλει αυτή η υπόθεση στην οικονομία. Και με αυτές τις οδηγίες θέλουμε να υλοποιηθεί η στρατηγική του 2020 και οι σχετικές δραστηριότητες και στόχοι. Οπότε αυτό το πρόγραμμα δράσης διαρθρώνεται ε, γύρω από τέσσερις ε, άξονες προτεραιοτήτων. Είναι οι βασικές προκλήσεις μας όσον αφορά τις ισχύουσες οδηγίες και ε, αυτές οι δράσεις μπορούν στο να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση, περισσότερη συνεκτικότητα και συνέπεια με τους στόχους μας που είναι κοινωνική και οικονομική. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ε, συμμόρφωση με τις οδηγίες, επίσης να έχουμε περισσότερες επενδύσεις για το Natura 2000 και να πάρουν περισσότερες συνέργειες. Επίσης οι κοινότητες και οι πολίτες να έχουν περισσότερη συνειδητοποίηση. 15 επιμέρους δράσεις προβλέπονται και σε αυτά τα δελτία τα οποία έχουμε δημοσιεύσει μπορείτε να δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες το χρονοδιάγραμμα αφορά τα έτη 2017 έως 2019. Θα τα πούμε και στις ερωταπαντήσεις που θα ακολουθήσουν, αλλά είπαμε ότι το πρόγραμμα δράσης δεν θα πρέπει να προθυκάσει το πώς θα διαμορφωθεί η νέα ΚΑΠ και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουν εμπλακεί επομένως στην Κομισιόν και η Επιτροπή των Περιφερειών η Τράπεζα Επενδύσεων, η Υπηρεσία για το Περιβάλλον. Να μην σας διαβάσω μία-μία τις δράσεις, αλλά για να δούμε τώρα όπως εδώ διατυπώνεται σε αυτές τις διαφάνειες ότι τα βασικά στοιχεία στην πρώτη δράση έχουμε το 1α και ένα β πώς, ε, για το οποίο θυμαθεί ο κ. Φλόρεντς, πώς θα μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε τις καυτήρες γραμμές και θα έχουμε κάποιους τομείς που θέλουμε να υπάρξει προστασία για σχέση με οικονομική δραστηριότητα και γι' αυτό ενδιαφέρονται οι κύριοι Χερμπράντι, η κυρία Μίλλερ και επίσης υπάρξουν κάποια άλλα μέτρα πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είδαμε τώρα Επίση, με αυτά τι καθημερινές γραμμέ τι θέλουμε να καλύψουμε. Είπε η Επιτροπή, το Σώμα των Επιτρόπων, τέλο πάντων, ότι θα πρέπει τα πράγματα να μείνουν ω έχουν, δεν θα θέλουμε να, αλήξουν, να αλλάξουν το κείμενο ή τα παραρτήματα. Και έτσι ε, θα πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση αυτών των κατευθυντηρίων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους και έτσι να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τις προσφερόμενες ευκαιρίες για τους μηχανισμούς ευελιξίας που υπάρχουν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ε, το άρθρο 6, 12 και 16 όσον αφορά τους κανόνες προστασίας των ειδών. Δεν μπορούμε, είπαμε, να προδικάσουμε το ε, τι θα προτείνει το κείμενο, τελικά θα ολοκληρωθεί με το 2018 και θα υπάρξει κάποια αξιολόγηση σε σχέση με τις σημερινές κατευθυντήριες και να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τον ε, έλεγχο επάρκειας. Έχουμε τις ε, εξαιρέσεις του άρθρου 16 και αυτό θα επικαιροποιηθεί και εκεί θα εξηγηθεί το τι ευελιξία μπορεί να δοθεί στο σημερινό πλαίσιο και να συζητήσουμε τις εθνικές αρχές με όλους τους εμπλεκόμενους και να ξεκαθαριστεί το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και ισχύουσα νομολογία. Σύμφωνα με αυτό τον έλεγχο της επάρκειας. Επίσης έχουμε τις οδηγίες για τα πτηνά και τους βιγότοπους και καλύπτουμε πάνω από 1.500 είδη. Ε, σε πάρα πολλέ περιπτώσει αυτό είναι προβληματικό λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, αλλά ακόμα και εκεί που υπάρχουν ε, προβλήματα και προστασία κάποιων ειδών και εκεί στις οδηγίες προβλέπεται κάποια ευελιξία και υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσεις για να μπορέσουμε να συγκεράσουμε τις διαφορετικές ανάγκες και αυτά επίσης καλύπτονται από τις κατευθυντήριες οπότε εάν είναι αποτελεσματικό αυτό το πρόγραμμα δράσης όσον αφορά το να μπορέσουμε να πετύχουμε στόχο της προστασίας τότε θα έχουμε ένα εργαλείο για καλύτερη χρήση της ευελιξίας στους μηχανισμούς προβλήματος. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα, τα συμβατικά σε σχέση με τα νομοθετικά προβλεπόμενα θα πρέπει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ό,τι μέτρα χρειάζονται για την προστασία. Να υπάρχουν ε, επί τούτου προγράμματα και τα κράτη-μέλη θα διαλέξουν τι είδου μέτρα χρειάζονται διοικητικά, νομοθετικά, συμβατική, σημαντικού χαρακτήρα. Τώρα έχουμε τη δράση 1B και λέει το πώς θα ενταχθούν αυτές οι υπηρεσίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, αυτό είχε απασχολήσει την κυρία Μπριάνο. ούτω ώστε να ενημερωθούν, να κινητοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι τα κράτη-μέλη για αυτές τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων, ούτω ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ισχύουσες πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουμε τα μαθήματα τα οποία μπορούμε να αντιλήσουμε από το τι ισχύει. Και αυτό να γίνει σε όλα τα επίπεδα στα κράτη-μέλη. Οπότε έτσι να υπάρξει χρηματοδότηση και μέσω της Eurostat και μέσω των δράσεων για το 2020. Έτσι αξιοποιηθεί η εμπειρία μας, ούτως ώστε αυτές οι υπηρεσίες να ε, ενταχθούν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και για όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσει κάποιες εκδηλώσεις όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συμμετάσχουν και έτσι όλοι να ωφεληθούμε από τα παραδείγματα προς μίμηση των κρατών μελών. Όλα αυτά θα είναι πολύ χρήσιμα. Για να δούμε τώρα τα θέματα που αφορούν τη δράση υπαριθμών 2. Να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον μηχανισμό υποστήριξης. Κάτι το οποίο είχε απασχολήσει τον κύριο Λίνς. Χρειάζονται και εδώ κατευθυντήρια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις αρμόδιες αρχές. Ούτως ώστε να υπάρξει μια ευφυής υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Γιατί όμως χρειάζεται ένα τέτοιο μηχανισμός. Γιατί το θέμα είναι η αδειοδοσία που προβλέπεται από τις ε, οδηγίες, από τις άριστες πρακτικές, ούτως ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμμετάσχουν και έτσι να ισχύσουν τα όσα περιγράφονται σε αυτά τα ενημερωτικά δελτία μας. Οπότε και ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν αυτόν τον μηχανισμό συνεννόησης των ομοτήμων Και έτσι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι άριστες πρακτικές και να συνεργαστούν οι εθνικές με τις περιφερειακές αρχές. Πάμε τώρα στην άλλη διαφάνεια. Έχουμε την επόμενη προτεραιότητα όσον αφορά την συμμόρφωση. Είμαστε στην δράση υπαριθμών 4, δηλαδή την ολοκλήρωση του Natura 2000 όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον και τα σχετικά μέτρα προστασίας και αυτό έχει απασχολήσει την κυρία Αγγιλέρα Γκαρθία. Και έχουμε τα σχετικά μέτρα, υποσχόμαστε για τη θάλασσα και άλλες δράσεις για να διευκολύνουμε τα μέτρα σε σχέση με την αλληλευτική πολιτική και να καλύψουμε τους ε, στόχους των σχετικών οδηγιών και την οδηγία πλαίσιο για τη θάλασσα και έτσι να έχουμε εύρυθμη λειτουργία των πολιτικών μας για τη θάλασσα και να υπάρχουν τα σχετικά μέτρα τα οποία καλύπτονται από τα πολιτικά προγράμματα για την αλία. Επίσης έχουμε κάποιες δράσεις για να διευκολύνουμε της, ε, της αφορμή των σχετικών ε, διεθνών συμφωνιών και διεθνών ε, οργανισμών και συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες τώρα. Έχουμε και κάποια άλλα μέτρα για, στις δράσεις 8, 9 και 11. Οπότε και εδώ έχουμε το θέμα την προστασία του περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση και ανταλλαγή αρίστων πρακτικών για να υπάρχει περισσότερη συνεκτικότητα ε, με τις δράσεις 6 και 13 στη θάλασσα έχουμε διαμερίσει συμφωνίες, συνεντήσει με τα κράτη-μέλη, οπότε και προκειμένου μπορούν να βοηθήσουν οι εμπλεκόμενοι και επίσης αναπτύσσουμε μεθοδολογία και κριτήρια για να μπορέσουμε περισσότερη συνεκτικότητα να προστατεύσουμε τη θάλασσα, το, το σχετικό δίκτυο σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και θεωρούμε ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν όσον αφορά το Natura 2000 στο κομμάτι που αφορά τη θάλασσα. Έχουμε τώρα τη δράση 6 και εδώ κάτι έχει ζητήσει η Αγγιλέρα Γκαρθία όσον αφορά την διασυνοριακή συμμόρφωση και εδώ να προσέξουμε ότι χρειάζεται αυτού του είδους η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και έτσι να φτάσουμε σε διασυνοριακή συμμόρφωση και σας υπενθυμίζω το ότι τα κράτη-μέλη έχουν αυτή την αρμοδιότητα και διασυνοριακά όσον αφορά την συμμόρφωση. Και τώρα για να δούμε κάποια άλλα ζητήματα σε σχέση με την δράση 7 όσον αφορά τα μεγάλα σαρκοφάγα ξάπλωσή του γιατί έχει ενδιαφερθεί αυτό ο κύριος Ντόρσμαν και η κυρία Μπριάνο. Και είπαμε να υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης για πολλά είδη από την αρμόδια ομάδα. Ε, αυτό είναι καυτό, επίκαιρο θέμα, τα μεγάλα σαρκοφάγα. Και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε ούτως είπε αυτά τα ζώα προς τις αργούδες, και να δούμε το πώς θα τα προστατεύσουμε αλλά στο φυσικό τους περιβάλλον. Και αυτό που έχουμε ως είναι ναι στην ε, επανεγκατάστασή τους αλλά αυτό είναι συμβατό με τις ανθρώπινες δραστηριότητες πάντως τα μεγάλα σαρκοφάγα είναι τμήμα της φύσης ε, και έχουν σημαντικό ρόλο για το περιβάλλον. Ο κόσμος έχει ξεχάσει πώς να αντιμετωπίσει το θέμα. Άρα θα πρέπει αυτή η γνώση να ξαναδιαδοθεί και να δούμε τι γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητε, ε, να δούμε τι θα γίνει με τους ε, λύκους που εξαπλώνονται και σε περιοχές όπου είχαν εξαφανιστεί για πολύ χρόνο. Αλλά όλα αυτά στη βάση της αρχής της ε, ενσωμάτωσης. Και οπότε και εμείς έτσι θέλουμε να ε, υπάρχει λιγότερη προστριβή και αντίθεση με τις ανθρώπινες δραστηριότητε. Οπότε έχουμε το πρόγραμμα live και άλλα προγράμματα για αναζήτηση λύσεων. Και έχουμε διάφορα προγράμματα λοιπόν, ούτω ώστε να υπάρχουν κάποια μέτρα συνύπαρξη και να μην υπάρχει πρόκληση ζημίας και συγκρούσει αντιθέτε. Προβλέπονται και αποζημιώσεις από αυτά τα σαρκοβόρα, εθνική πόρη είναι αυτό και επίσης κάποια μέτρα πρόληψης, διάφορα μέτρα, ηλεκτροφόρα καλώδια, ε, προστασία με σκύλους και για τις αρκούδες τεχνική αρρωγή, για διάφορους ε, μπλεκόμενους, διάφορες εκστρατείες, ε, ομάδες που βοηθούν, ας πούμε όσον αφορά τις προβληματικές αρκούδες που πολλές φορές έχουν επικίνδυνη συμπεριφορά κατά των ανθρώπων. Και όταν δεν υπάρχουν ικανοποιητικέ εναλλακτικέ, έχουμε κάποιες παρεκκλήσεις, οπότε επιτρέπεται η εχμαλωσία, η παγίδευση τέλο πάντων προστατευομένων ειδών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη όπου υπάρχει, υπάρχουν πρακτικές ε, αρμονικής συνύπαρξης οπότε έχουμε και αυτή την πλατφόρμα για την συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων και για να δούμε τώρα το άλλο θέμα τι γίνεται με την ομάδα συντονισμού για τα πουλιά Αυτά θεσπίζονται ε, σε κάποιο πρόγραμμα του live. Έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και έχουμε 5 με 7 μέλη σε εβδομάδα συντονισμού για το live. Ε, και οι φορείς των κυνηγών, όχι όμως τα κρατη Πάντως θα υπάρξει κάποιος μηχανισμός που θα εξασφαλίσει την συμμετοχή των κρατών μελών όταν έρθει η ώρα να ρυθμίσουμε τις πρακτικές λεπτομέρειες και τον ρόλο αυτού του μηχανισμού συντονισμού στα πλαίσια του LIFE. Αλλά καταρχήν θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα αυτή η ομάδα, θα τεθούν και προτεραιότητες, ποια πουλιά χρειάζονται ε, προστασία, πλαισίωση και να δούμε τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη από πλευρά του. Και τώρα, για να δούμε την προτεραιότητα C. Για τις επενδύσεις και μετά θα έρθω σε κάποια θέματα επενδύσεων. Όπως ε, παραδείγματο χάρη με τις ερωτήσεις του κύριου Φλόρεν, της κυρίας Κάντενμπαχ, για τις λήψεις ε, της χρηματοδότησης ε, που δεν έχουν αντιμετωπιστεί καλύτερα στο σχέδιο δράσης. Επίσης υπάρχει η ερώτηση της κυρίας Καμπεσόν Ρουής για την αποζημίωση γεωκτημόνων, τα παρελθόντα μαθήματα, σύνδεση με άλλα ταμεία, μελλοντικέ χρηματοδοτικές απαιτήσει από τον κύριο Ντεμέσμακερ και επίσης την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων επίσης από τον κύριο Ντεμέσμακερ. Θα ξεκινήσω με το εξής. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, το σχέδιο δράσης έχει στόχο να προωθήσει την εφαρμογή των οδηγιών βραχυπρόθεσμα, δηλαδή 2017-19 με το υφτάμενο νομικό πλαίσιο και πι δέλτα πι. Ε, βεβαίως να προωθήσει και διάφορες μεταρρυθμίσεις της κοινή γεωρικής πολιτικής στο σχέδιο δράσης αυτό. Οπότε βεβαίως γνωρίζουμε όλοι τις ελλείψεις ε, χρηματοδότησης ε, που προκύπτουν είναι ένας παράγον κλειδί που εμποδίζει την καλύτερη εφαρμογή και αυτά θα αντιμετωπιστούν για την περίοδο 2017-19. Θα βρείτε τις δράσεις 9-10-11, 9 και 10 αφορούν την κυνηγιορική πολιτική και η 11 αφορά το Ταμείο Αλίας όπου προωθούμε μέτρα για την καλύτερη χρήση μεταξύ των οποίων στα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου να προωθούμε καλύτερα τέτοια συστήματα. Τώρα το σχέδιο δράσης έρχεται με, έχει την μορφή βελτίωσης ε, του οικονομικού σχεδιασμού για το Natura 2000. Ε, δηλαδή τα σχέδια ε, δράσης κατά προτεραιότητα τα σχέδια αυτά, δηλαδή για το 17, 18, 19, θα είμαστε έτσι σε θέση να γνωρίζουμε καλύτερα για το επόμενο πι δελτα πι, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών. Το θέμα της ε, αποζημίωσης. Η αποζημίωση για τους γεωκτήμονες βεβαίω υπάρχει ως δυνατότητα ήδη σήμερα στην κυνηγυρική πολιτική. Στην δράση 9 η Κομισιόν θα ενθαρρύνει την πλήρη και αποτελεσματική χρήση των πόρων για το, τους χώρους Natura 2000. Θα προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε και να προωθήσουμε γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτό πιο συχνά γιατί δεν το εκμεταλλεύονται τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε να βελτιωθεί η κατάσταση μέχρι το 2019 για την παρακολούθηση των ε, ταμείων για την βιοπικιλότητα. Υπάρχει μια σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου προς την Κομισιόν για να υπάρξουν οριζόντι δείκτες για το Natura 2000 για όλα τα ταμεία και θα δούμε τους υφιστάμενους δείκτες και τη δυνατότητα να φτιάξουμε νέους δείκτες όπου αυτό είναι δυνατόν χωρίς να προδικάζουμε αυτή τη στιγμή τις συζητήσεις για το επόμενο πι δελτα πι. Τώρα, Αυτά αφορούσαν τις γενικές ερωτήσεις για την προτεραιότητα. Τώρα για την δράση 8. Υπήρχε μία ερώτηση της κυρίας Αγγιλέρα Γκαρσία, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την συνέργεια μεταξύ Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και του ιδιωτικού τομέα επαρκώς ε, ή από τον κύριο Μάκερ, αν σκοπεύουμε να έχουμε περαιτέρω συγκεκριμένα κριτήρια για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το οποίο βρήκαμε είναι ότι υπάρχουν σήμερα αρκετά καινοτόμα εργαλεία για να προωθήσουμε την προστασία από ιδιώτες που υπάρχει ήδη και συμβαίνει στην Ευρώπη και αλλού, ειδικά στις ΗΠΑ και σκοπεύουμε να τονώσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις στην προστασία της φύσης, ε, στηρίζοντας έργα που στόχο έχουν την ενίσχυση ιδιωτών και ιδιωτικών οργανώσεων. Πρόκειται για μια εθελοντική προσέγγιση προστασίας ιδιωτικής γης. Δεν βλέπουμε ε, πέρα κανένα πρόβλημα. Πράγματι μπορεί να υπάρξει συνέργεια με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα για το χρηματοδοτικό μέσο για την ε, προστασία της φύσης. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις αυτές είναι επιλέξιμες μόνο όταν συνεισφέρουν στη βιοπικιλότητα και την ε, προσαρμογή στην ε, κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τον κανονισμό LIFE. Οπότε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση τη συνεισφορά ε, του κάθε έργου σε αυτούς τους στόχου και αυτό πρέπει να το λάβει μετά υπόψη η όταν αξιολογεί την επιλεξιμότητα του έργου. Και επιπλέον οι επενδυτές που λαμβάνουν την ε, χρηματοδότηση θα πρέπει να παρακολουθούν το αποτέλεσμα που υπάρχει όσον αφορά την προσαρμογή και τον αντίκτυπο. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε επαρκή κριτήρια. Περνάω στην ερώτηση 9 που αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Το ερώτημα ήταν εάν εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε κάποια αξιολόγηση, αυτό το οποίο έθεσε ο κύριος Λόρεντς, επίσης ερώτημα για περαιτέρω λεπτομέρειες και συνέργεια με την ΚΑΠ που έθεσε η κυρία Γκαρσία και επίσης αν είναι αρκετά φιλόδοξο το σχέδιο δράσης ε, του κυρίου Γκερμπράντη ερώτηση για την αξιολόγηση στην ε, βιοπικιλότητα και στην χρήση οικονομικών πόρων για βιοπικιλότητα και Natura 2000 ε, και για την χρήση των μέτρων Natura 2000 για να αντισταθμίσουμε ε, τα, της αλληλείας, ε, τα διαφυγόντα κέρδη. Αυτό θα γίνει με μία ξεχωριστή μελέτη. Οπότε ο στόχος είναι να αξιολογήσουμε το ποσό των χρημάτων ε, που ξοδεύεται και πώς αυτό γίνεται. Και ποια αποτελέσματα θα επιτύχουμε. Για την αποζημίωση τώρα, ο λόγος για τον οποίο το αναφέρουμε είναι ότι έχουμε την ε, αίσθηση ότι αυτό δεν ε, έχει χρησιμοποιηθεί επαρκώς και υπάρχουν έτσι εντάσεις με τους αγρότες. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης χρήσης ε, για να μην υπάρχουν ακριβώς αυτές οι αντιδράσεις αν υιοθετηθεί περαιτέρω. σημαντικό είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αξιολογήσουν την υφιστάμενη χρήση των κονδυλίων και να φροντίσουν οι αγροπεριβαλλοντικές αρχές να μοιραστούν την ευθύνη για την διαχείριση των εκτάσεων το 2000 με τους αγρότες και να εκπαιδεύσουν τους αγρότες μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κάτι το σημαντικό, εάν μου επιτρέπετε για την κοινή γεωργική πολιτική, είναι το ότι υπάρχει μία μείωση των ειδών και των ενδιαιτημάτων που ζητάει βεβαίως μια μεγαλύτερη, απαιτεί μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση των και των κονδυλίων. Οπότε η πρόταση της Κομισιόν για να απαγορευτεί η χρήση ζυζανιοκτώνων σε περιοχές οικολογικής έμφασης εγκρίθηκε από την ε, Επιτροπή Γεωργίας και ελπίζω να εγκριθεί και από την Ολομέλεια. Ε, οι περιοχές αυτές αφορούν την βιοπικιλότητα επίσης και έχει νόημα νομίζω και να απαγορευθούν ακριβώς ε, τα ζητανιοκτώνα. Τώρα θα περάσουμε ερώτηση 11 βασικούς οικονομικούς τελεστές όπως είναι αλληλείς, κάποιες οργανώσεις, ε, πόροι για βιώσιμους αλληλευτικούς τρόπους και τα ωφέλη ε, προς τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα του, της Ελίας ως ε, τομέα που θα εξασφαλίσει τη διασφάλιση και των οικοσυστημάτων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ανάμειξη και των ελίων και των οργανώσεών τους ε, και οργανώσεων για την προστασία των ε, θαλάσσιων και αλληλευτικών πόρων. Είναι σημαντικοί φορείς και τελεστές και θα ε, αναπτύξουμε έτσι και κάποια νέα μέτρα στα πλαίσια την κοινή αλληλευτική πολιτική για, τα, για τις περιοχές θαλάσσιες, για θαλάσσιες περιοχές των Natura 2000. Και με τη δράση 11, διευκολύνοντας την καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων που έχουμε για τη βιοπικιλότητα, μπορούμε να προωθήσουμε ε, τα θέματα αυτά και στην Αλία. Τώρα, οικοτουρισμός, οικολογικός τουρισμός και βιώσιμη αλία. Σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων σε προστατευμένες θα, θαλάσσιες περιοχές. Μία συναφής ερώτηση προς τη δράση 12. Είναι η ερώτηση του κ. Μερσμάκερ για τη χρηματοδότηση της συνδεσιμότητας των πράσινων υποδομών μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων. Έχουμε καταρχήν μια δράση που στόχο έχει την ανάπτυξη κριτηρίων για πανευρωπαϊκές οικολογικές υποδομές που μπορεί να περιληφθεί και στο επόμενο ΠΔΠ και στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για να βελτιώσουμε την τρέχουσα χρήση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τους πόρους ε, για τις οικολογικές υποδομές. Πάντως, επαναλαμβάνω, έχουμε και τη διαβλό των, της αγροτικής ανάπτυξης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση για την ε, ευρύτερη ανάμειξη, ρώτησε Μπριάνο και πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει στην εξάπλωση και διάδοση των δράσεων προκειμένου να αποφέρουν καρπούς. Το σχέδιο δράσης είναι για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ε, και φυσικά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό ε, έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρόλο για την μετάδοση του σχεδίου αυτού, για την πρόθεση καλών ε, πρακτικών και ανέβρεση λύσεων και την εμπλοκή περισσότερων ε, ενδιαφερομένων, κυρίως ε, γεωκτημόνων. Ε, έχουμε μάλιστα μεταφράσει το έντυπό μας σε όλες τις γλώσσες, ώστε μπορείτε να το προωθήσετε και σε εκλογικές περιφέρειες, στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη η ανάμειξη και το. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι δράσει που έχουν προστιθέμενη αξία για τις συζητήσεις στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι πολύ σημαντικό και στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά το σημείο 13. Ερώτηση Μπριάνου για το πώς θα εμπλέξουμε καλύτερα την Επιτροπή των Περιφερειών, πώς θα ληφθούν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις της και επίση τεχνική πλατφόρμα για περιβαλλοντική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Περιφερειών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας διαβεβαιώ ότι το σχέδιο δράση λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών που συμμετείχε ήδη στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσεως και δράσεις όπως η 161314 13-14 δεν θα κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πόρους θα αφιερώσει η Επιτροπή των Περιφερειών στα θέματα αυτά. Πάντως είμαστε πεπισμένοι ότι ε, αναμειγνύεται πλήρως ε, στην εφαρμογή του σχεδίου δράσεως και η Επιτροπή Περιφερειών. Σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα για τη συνεργασία, την περιβαλλοντική συνεργασία, ήδη λαμβάνει η χώρα, θα ε, πολλαπλασιαστούν όμως τα εργαστήρια, τα σεμινάρια, οι διασκέψεις για να προωθήσουμε την ε, καλύτερη και σπευσμένη εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Αναφέρεται και στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που σύστησαν η Επιτροπή Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολυνθεί ο διάλογος και η κοινή χρήση πληροφοριών προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της, νομοθεσία στο τοπικό επίπεδο. Και φυσικά ε, ισχύει κάτι τέτοιο και στις οδηγίες για τη φύση. Η κυρία Μπριάνο έθεσε μια ερώτηση για τη δράση 14 για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και κατά πόσο καλύπτεται από τη σχετική δράση, την 14 και πώς μπορούν οι πολίτες ε, να ε, συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που είναι το 2018. Καταρχήν και η ηλική και άλλη πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ε, καλύπτεται στη δράση 14. Και επίσης συνέργειες μεταξύ των άλλων πολιτιστικών αγαθών και φυσικών οικοσυστημάτων λαμβάνονται υπόψη για να ενισχύσουμε αυτή τη συνέργεια μεταξύ των δύο πτυχών της κληρονομιάς μας και η συμμετοχή στη στο ε, Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς ε, ήδη δρομολογείται από όλα τα θεσμικά όργανα και ήδη συνεργαζόμαστε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εθνικούς φορείς για ε, προγράμματα όπως το πρόγραμμα για την Δημιουργική Ευρώπη. Ποια είναι τα μελλοντικά βήματα. Φυσικά, το σχέδιο δράση είναι πολύ φιλόδοξο, με την εμπλοκή πολλών παραγόντων ε, για τα μισή χρόνια. Ήδη υπάρχουν και, και η ανακήρυξη της ε, ημέρας για το Natura 2000. Έχουμε διάσκεψη στις 6, διάσκεψη στις 6 Ιουνίου κοινή διοργάνωση με τη Μαλτέζικη Προεδρία και την Επιτροπή Περιφερειών, όπου ο αντιπρόεδρο Τίμερμαν διατράνωσε τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το περιβάλλον και τη φύση και το σχετικό σχέδιο δράση. Και μάλιστα περιμένουμε και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου. Έγιναν όμω κάποιε γενικέ ερωτήσει για το σχέδιο δράση. Δεν ξέρω αν έχουμε αρκετό χρόνο για να απαντήσω. Καταρχήν είχαμε μία ερώτηση του κυρίου Πότς που ρώτησε γιατί δεν δώσαμε περισσότερη έμφαση σε, σε συγκεκριμένους τομείς, σε γεωργία, μεταφορές, ενέργεια που επηρεάζουν ιδιαίτερα το περιβάλλον. Φυσικά όλες οι δραστηριότητες ε, επηρεάζουν το περιβάλλον, γι' αυτό προτιμήσαμε να μην ε, διαχωρίσουμε τους διάφορους κλάδους, αλλά να συμπεριλάβουμε γενικά τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χωρίς διαχωρισμό ανακλάδο. Πιστεύουμε ότι έτσι θα είναι καλύτερη η προσφορά. Επίσης, ε, γιατί δεν λάβαμε υπόψη και τα έντομα επικονίασης, ρώτησαν οι κύριοι Πότστε, Μαρσμέκερ και Μπέαρντερ. Ναι, γνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα έντομα επικονίασης έχουν κέριο ρόλο στην φύση και στην οικονομία. Και είναι σημαντική υπηρεσία οικοσυστήματος που ε, παρακμάζει δυστυχώς. Και πολλά είδη εντόμων επικονίασης και άλλων ε, ειδών επικονίασης λαμβάνονται υπόψη στην νομοθεσία για τη φύση. Αλλά θεωρούμε ότι το θέμα είναι ευρύτερο. Αφορά τη γεωργία, την υγεία των φυτών, την έρευνα. Δεν είναι μόνο θέμα των φορέων της επικονίασης. Οπότε το θέμα αυτό της επικονίασης θα το λάβουμε υπόψη, αλλά όχι συγκεκριμένα εντός του σχεδίου δράσεως. Επίσης, ρωτήθηκε για δεν είχαμε μια πρωτοβουλία για τις πράσινες υποδομές ε, σε διευρωπαϊκό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μια δράση που προωθεί τις πανευρωπαϊκές οικολογικές υποδομές ε, ε, με αποκατάσταση και διασυνδεσιμότητα των περιοχών της Natura 2000. Δεν θέλουμε να προεξοφλήσουμε καμία πτυχή του επόμενου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και τα κριτήρια των υποδομών ίσως συμπεριληφθούν στη συνέχεια στο ΠΔΠ αν ε, χρειαστούν συγκεκριμένες δράσεις ε, διευρωπαϊκών δικτύων. Ε, οπότε με τις καταθυντήριες γραμμές που θα λάβουμε θα δούμε πώς θα προσδιορίσουμε κάποιες σημαντικές πανευρωπαϊκές πράσινες υποδομές για να συμπεριληφθούν αργότερα στο ΠΔΠ. Επίση, ε, για τη στρατηγική βιοπικιλότητα, ερωτήσεις Δεμεσμέκερ και Γερπράντη. Σίγουρα το σχέδιο δράση θα συμβάλλει σημαντικά στο, στην υλοποίηση του στόχου βιοπικιλότητας. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι από μόνο του το σχέδιο δράση δεν, δεν μπορεί να μα εξασφαλίσει την υλοποίηση των στόχων βιοπικιλότητας. Χρειάζονται και άλλε δράσει που ξεπερνούν τι οδηγίες για τη φύση. Για παράδειγμα, οι στόχοι 2, 3, 5 και 6 ε, δεν, φαίνεται ότι μόνο του το σχέδιο δράση δεν είναι πανάκια για την υλοποίηση της βιοπικιλότητας. Τώρα θα συγκεντρωθεί η πολιτική βούληση για την υλοποίηση των στόχων βιοπικιλότητας. Θα δοθεί περισσότερη προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, όπως είπα, ε, απαρτίζεται από 15 συγκεκριμένες δράσεις και 100 δευτερεύουσες δράσεις. Ε, θα εγκαινιαστεί το 2017 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2018. Προσβλέπουμε σε ε, εσπευσμένη εφαρμογή και, και το σχέδιο δράση και οδηγίες για τη φύση είναι στέρα θεμέλια για την προώθηση της βιοποικιλότητας. Χρειάζεται όμως μια πολιτική βούληση και υποστήριξη και με υπόψη το σχέδιο δράσης. Δεν ήταν μόνο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς, ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν και πολλές υπηρεσίες και διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ήταν μοναδικό προνόμιο της ε, Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Φαίνεται λοιπόν από αυτή τη συλλογική δράση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσιλωμένη στο θέμα αυτό και ευελπιστούμε ότι την ίδια δέσμευση, στράτευση και πολιτική βούληση θα την επιδείξουν και τα κράτη-μέλη. Τώρα, θα λάβει το, το σχέδιο δράση υπόψη την ιδιαιτερότητα των κρατών μελών, ρώτησε ο κύριο Γκερπράντη. Ε, τα κράτη-μέλη φυσικά λαμβάνονται υπόψη στις διαβουλεύσεις και μέσω των διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων και Γι' αυτό έχουμε και διμερείς διαλόγους με τα κράτη-μέλη, έχουμε μπλέξει και την Επιτροπή των Περιφερειών για να λάβουμε υπόψη και το τοπικό και περιφερειακό παράγοντα, οπότε λαμβάνονται έτσι υπόψη ιδιαιτερότητες οι εθνικές. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των κρατών και των ενδιαφερομένων. Όταν έγινε ο έλεγχο καταλληλότητα, έγινε και με συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των κρατών μελών. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το σχέδιο δράσης λαμβάνει υπόψη αυτές οι ιδιαιτερότητες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη δεν θα, θα συμμετέχουν επαρκώς. Τώρα, γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν κάποιες συγκεκριμένες δράσεις στο σχέδιο δράσης. Ο κύριος Γκερμπράντι ανέφερε το ζήτημα το προστατευμένο δράσος Μπιελοβιέζα στην Πολωνία και μας είπε αν μπορούμε να ενημερώσουμε για την ε, υλοτόμηση που γίνεται στο δάσος αυτό. Οι πολωνικές αρχές έδωσαν μια απάντηση στην ιτιολογημένη ε, γνωμοδότησή μας για την υλοτόμηση στο δάσος Μπιελοβιέζα και οι πολωνικές αρχές ε, κατέριψαν ε, την ε, δήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καταστρατήγηση της οδηγίας ε, Natura 2000 και πιστεύουμε ότι δεν θα σταματήσει η λοτόμηση δυστυχώς στο δάσος Μπιλοβέζα αφού αναλύσουμε διεξοδικά τις απαντήσεις πολωνικής κυβέρνησης που καταρρύπτει τις κατηγορίες για καταστρατήγηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θα δούμε κατά πόσο θα ασκήσουμε προσφυγή εις βάρος της Πολωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα όσον αφορά τους χορτολιβαθικές ε, εκτάσεις, Α, ήταν κάποια άλλη ερώτηση επομένω και το θέμα κατά πόσο μπορεί να γίνει αποχαρακτηρισμό και είπαμε ναι ότι αυτό τεχνικά γίνεται. Είναι θέμα σημαντικό για το περιβάλλον, αλλά όμως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτό, ειδικέ περιπτώσεις, να για παράδειγμα, εάν από πλευρά περιβάλλοντος ε, ο αποχαιρετισμός θα, θα ωφελούσε και αυτό περιέχεται στο κάποιο έγγραφό μας όσον αφορά την κάποια το περιβάλλον. Και είπαμε ότι στο Natura 2000 θα πρέπει να υπάρξει μόνιμος χαρακτηρισμός τέτοιων χορδολιβαδικών εκτάσεων και έχουμε, είπαμε, κάποια τέτοια δράση που θα προωθεί αυτό τον στόχο. Έκανα ό,τι μπορούσα για να απαντήσω τις ερωτήσεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για αυτή την τόσο εξαντλητική πλήρη σας εισήγηση. Αλλά έτσι έπρεπε να γίνει γιατί 45 ήταν οι βουλευτές που άψασαν απίφθηναν ερωτήσεις. Φαντάζομαι ότι έχουν καλυφθεί. Οι συνάδελφοι παρόλα αυτά, όποιος θέλει μπορεί να ζήσει το λόγο για κάποιο είδου επερώτηση, σχόλιο. Ο κύριος Φλόρενς και ο κύριος Ντόρφμαν έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Κάντεμπαχ επίσης. Σίγουρα θέλει το λόγο ο Ντεμές Μάκερ και θα έχουμε και δεύτερο γύρο ερώτα απαντήσεων για τους συναδέλφους που δεν είχαν υποβάλει αρχικά ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο κύριο Φλόρενς. Από ό,τι βλέπω, δουλέψατε πάρα πολύ. Καλά κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας, ούτως ώστε να υπάρξει αίσια συνέχεια για το Natura 2000. Και ως Γεωργός και εγώ επίσης έπρεπε να εφαρμόσω ό,τι προβλέπετε και άλλα να σας τα πω με ειλικρίνεια. Δεν έχω πρόβλημα με το Natura 2000. Ό,τι το να πάθω, το έπαθα τέλος πάντων. Οπότε τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που μας προβληματίζουν. Για παράδειγμα, τι είναι με τους κορμοράνους ή τι θα γίνει με τους λύκους. Και στη Γερμανία αλλά και στην Αυστρία ε, πρόκειτο για τραγωδία, για καταστροφή. υπήρχε επαρκές αξιόλογο επίπεδο προστασίας των ειδών αυτών. Και ε, πάντως όποτε κάποιοι κυνηγοί στράφηκαν αντίον αυτών των ειδών, αμέσως παρενέβησαν μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους έσυραν στα δικαστήρια. Είναι θέμα διακομματικό αυτό. Όμως θα πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εξωθεί στην ανεργία ένα σωρό ψαράδες διότι θα, θα χάσουν τη δουλειά τους εάν κατά λάθο εχμαλωτήσουν, πιάσουν τέλος πάντων, ψαρέψουν έναν κορμοράνο. Η Σουηδία έχει σοβαρά με το θέμα των θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανασταθμίσει αυτά τα οποία έχει θεσπίσει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές προστρεβές μεταξύ Σουηδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επιτροπής. Και επίσης ξέρουμε ότι οι λύκοι στη Σουηδία έχουν στραφεί κατά ταράνδων ε, και ελαφιών. Και λόγω των λύκων σκορπίζονται τα κοπάδια των κτηνοτρόφων και δεν μπορεί και να ξαναμαζέψουν τα ζώα τους. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη με τους λύκους. Θα πρέπει επομένως να δοθεί μία λύση. Δεν λέμε ότι πρέπει η Επιτροπή να ικανοποιήσει κάθε αίτημα των Γεωργών. Εντάξει, στη Γερμανία δεν είμαστε και στη χειρότερη κατάσταση αλλά δεν ξέρω εάν οι αποζημιώσεις που προβλέπονται πρόκειται να φέρουν, να οδηγήσουν τέλο πάντων τους κτηνοτρόφους στο να φυσικάσουν και να μην κυνηγούν τους λύκου. Υπολείπονται πολύ αυτές οι αποζημιώσει από το τι θέλουν οι κτηνοτρόφοι. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σήμερα δεν αναφέρθηκε καθόλου το ότι θα πρέπει να έχουν οι ασχολούμενοι με τη γεωργία ένα εισόδημα που τους εξασφαλίζει τα ζήν. Και εγώ είμαι γεωργός. Ναι, να εφαρμοστούν τα σχετικά μέτρα, αλλά να υπάρχει και κάποιο εισόδημα. Επί τρία έτη το γάλα ήταν πιο φτηνό από το νερό. Ε, πώς να ζήσει έτσι ένας Γιώργος. Δεν θέλω να υπονομεύσω τα προγράμματά σας, αλλά καθίστε και επαναξιολογήστε την ΚΑΠ. Γιατί προς το παρόν είναι τουλάχιστον μια παραδοξότητα. Ευχαριστούμε κύριε Φλόρεντς. Ο κύριος Ντόρφμαν είναι ο επόμενος που το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. συνεχίσω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φλόρεντς. Ναι, όσον αφορά τη σχετική οδηγία και τα της προστασίας των ειδών, ότι θεωρητικά τα λέει καλά. Όμως, στην πράξη τα είπε ο κ. Λόρεντς σε σχέση με τους λύκους και άλλα είδη. Πρόκειται για είδη που σε ε, πολλά μέρη της Ευρώπης απειλούνται με εξαφάνιση. Έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες. Αλλά υπερακοντίζουν τον στόχο μας. Θα πρέπει επομένω, είπαμε, να υπάρχει ευελιξία. Που υπάρχει, αλλά μόνο στα χαρτιά. Ρίξτε μια ματιά στο πόσα ήδη έχουν ή δεν έχουν μάλλον επαναξιολογηθεί και επανακαταταχθεί. Τα τελευταία χρονιά, είπαμε τι γίνεται με τους λύκους, τα είπαμε και στην Επιτροπή των Περιφερειών τις προάλλες τι γίνεται όσον αφορά τη συνύπαρξη ανθρώπων και λύκων, ε, τι γίνεται σε σχέση με την ορεινή γεωργία, τι γίνεται με τις χορτολεβαδικές ε, εκτάσεις, Δηλαδή, είναι κάτι σαν τις πόλεις ε, όπου συμβιούν οι άνθρωποι με τους αρουραίους, δηλαδή ότι ναι, συμβιούν, αλλά τα πράγματα είναι προβληματικά. Αυτό ισχύει και για τους λύκους. Άρα, είδαμε ότι σε τρία χρόνια διπλασιάστηκε σε πολλές χώρες ο πληθυσμός των ε, ε, λύκων, χρειάζεται μια φυσική ισορροπία και αυτό Ε, δεν μπορεί να οδηγεί στο να αποδεκατίζουν οι λύκοι έγιες και πρόβατα. Και στη περιοχή έχουμε εγώ πρόβατα. Οπότε τι θα γίνει, θα υπάρχει προστασία των λύκων ή θα υπάρχει προστασία των εγωπροβάτων. Και στην Ιταλία υπάρχουν χιλιάδες λύκων. Και πολλές φορές διασταυρώνται και με τους σκύλους. Και δεν είναι συχνά ο κέντρο ευρωπαϊκός λύκος εκεί, αλλά ένας υβριδικός πληθυσμός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, γιατί δεν μιλάμε πλέον για προστασία του συγκεκριμένου είδους. Σε λίγα χρόνια στην Ιταλία θα έχουμε μόνο το υβριδικό αυτό είδος. Γιατί διασταυρώνονται με σκυλιά πάρα πολύ εύκολα οι λύκοι και έχουμε όπως σας είπα αυτό το υβρίδιο, το υβριδικό είδος. Τι σημαίνει αυτό. Τι είναι το λογικό και ποια είναι η λογική συνύπαρξη μεταξύ της αναγκαιότητας ε, της γεωργίας και της ορεινής ε, γεωργίας και της βιοπικιλότητας και τι θα επιτύχουμε με τον ε, και πόση περισσότερη βιοπικιλότητα θα έχουμε ή λιγότερη βιοπικιλότητα αν θέλετε γιατί αν εξαφανιστεί η ορεινή γεωργία και εκτινοτροφία δεν ξέρω εάν αυξηθεί όντως η βιοπικιλότητα ή απλά θα έχουμε μια αύξηση των ή ιδνίων των των λύκων. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κάντενμπαχ. ιδιων των λυκων πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση και την απάντηση των ερωτήσεών μας. Πάρα πολύ καλή δομή. Μια συμπλήρωση Λυπούμε για το ότι κάποια μέτρα δεν βρήκαν ανταπόκριση όπως περιγράψατε. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να το δούμε αργότερα. Το τρίτον σχετίζεται με αυτό το οποίο είπε ο προλαλής σας. Ε, δεν συμφωνώ με όλα όσα είπε, αλλά με αρκετά. Είχαμε τότε τη μεγάλη συζήτηση με τον Κάστορα, τώρα έχουμε τη μεγάλη συζήτηση με τα ψάρια. Δηλαδή το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να εξαφανιστεί, δεν είναι μόνο οικονομικό δε το ζήτημα, αλλά είναι και θέμα αποδοχής των περιοχών 2000 γιατί βεβαίως ε, αυτοί οι οποίοι θίγονται, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί έχουν πολύ ισχυρά λόμπι και στα ΜΜΕ. Από την άλλη έχουμε την προστασία της, φύλης, ε, της φύσης. Θεωρώ λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση αν θέλετε, σε μια κατάσταση ε, που συχνά υπάρχει χωρίς ε, να υπάρχει επιστημονική θεμελίωση. Και ε, αυτό νομίζω θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με πιο ξεκάθαρες αποφάσεις και διατάξεις από πλευράς Κομισιών Γιατί τώρα βλέπουμε πίεση της κοινή γνώμης και τελικά καταλήγουμε πάντα σε μισές λύσεις. Αν αναφέρουμε τα παραθυράκια να αναφέρουμε την πολύ ελαστική ερμηνεία των διαφόρων ε, διατάξεων. Π.χ. έχουμε μια περιοχή και μετά έχουμε κάποιες εξαιρέσεις μέσα στην περιοχή, γεωγραφικές δηλαδή. Τότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχουμε ξεκάθαρες λύσεις και αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως πάντα όλα τα συμφέροντα, χωρίς όμως ε, παραθυράκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την ε, Κομισιόν για την πολύ καλή παρουσίαση και απαντήσεις και εκτιμώ πραγματικά τον κόπο που έκαναν ε, για να απαντήσουν. Βεβαίω έχουν μείνει κάποια ζητήματα να πάρουν. Αλλά να πω πρώτα απ' όλα ότι περιμένουμε πάρα πολλά από αυτό το σχέδιο δράσης ε, οπωσδήποτε μια καλύτερη κατεύθυνση για την ε, εφαρμογή που πρέπει να βελτιωθεί η πραγματική εφαρμογή επιτόπου. Και εδώ πέρα βεβαίως κοιτάει στο μέλλον το σχέδιο δράσης, αλλά βεβαίως ε, το θέμα είναι να επιτύχουμε τους στόχους της βιοπικιλότητας 2020 και εκεί πέρα η Κομισιόν παραδέχεται ότι θα απαιτηθούν κάποια περισσότερα πράγματα. Ότι αυτό δεν αρκεί δηλαδή και ε, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς η Κομισιόν θα προωθήσει κάτι τέτοιο και ποιο είναι το σχέδιο επίσης μετά το 2020. Πρόκειται για ένα πρόβλημα ε, το οποίο εξορισμού απαιτεί ένα όραμα πιο μακροπρόθεσμο, μια δράση πιο μακροπρόθεσμη, ενώ εμείς δρούμε με κάποια πλαίσια τα οποία είναι σχετικά βραχυπρόθεσμα. Ε, είναι κάποιο μειονέκτημα αυτό, αλλά τελικά το όραμά μας, ε, η πράξη μας θα πρέπει να διαμορφωθούν κάπως πιο μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό έχω προτείνει και κάποιες δράσεις ε, στην έκθεσή μου. Να που αφορούν παραδείγματος χάρη τις πράσινες υποδομές, ε, το δίκτυο TNG, όπου ε, πραγματικά εκεί πέρα δεν υπάρχει μια πραγματική συγκεκριμένη πρόταση. Εντάξει, έχουμε μπλέξει στα, στα άμεσα, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε κάπως καλύτερα το μέλλον. Να έχουμε καλύτερες συνδέσεις, πράσινη υποδομή. Το ίδιο επίσης ε, για το πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε ε, των διαχειριστών ε, που επίσης αναβλήθηκε αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και εδώ πέρα αναμένω από σας περισσότερη συνέπεια και όραμα για το τι θα πρέπει να γίνει μακροπρόθεσμα. Οπότε θέλω να παρακυλήσω την Κομισιόν να ρίξει εκεί το βάρος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκαν. Σας ευχαριστώ. Κατά τη γνώμη, κατά την εμπειρία μου, το πιο σημαντικό θέμα για τις οδηγίες για τα πτηνά και τα αντιτήματα, το πιο σημαντικό θέμα είναι η επικοινωνία. Και συμφωνώ με την διατήρηση, είναι πολύ σημαντικό και το μέλλον μας εξαρτάται από αυτή. Αλλά χωρίς διαβουλεύσεις έγκαιρες, τότε θα πάνε όλα στραβά. Και σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα διατήματα των πτηνών, στην Ιρλανδία δεν είχαμε διαβουλεύσεις. Ουσιαστικά μας παραγωνίσετε, ε, χαρακτηρίστηκαν ε, περιοχές Natura 2000 χωρίς καμία διαβούλευση, μάλλον για τα αντιτήματα ε, για τα πτηνά, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία. Απλώς λάβαμε ενημέρωση, κοινοποίηση ότι οι... τα εδάφη χαρακτηρίστηκαν. Και μάλιστα ε, για 600 χρόνια είχαμε συγκεκριμένες ονομασίες και δεν δόθηκαν καν συγκεκριμένες ονομασίες για το χαρακτηρισμό των εδαφών. Για παράδειγμα, εγώ αγοράζω τα κάψιμά μου από κάποιο που λέγεται Club Chambers Bag. Clunking Bag εμεί τη λέγαμε αυτή την περιοχή για χρόνια ολόκληρα, για εκατοντάδε χρόνια. Τώρα αν πείτε σε κάποιους ότι σε συγκεκριμένο αγροτεμάχη δεν μπορούν να κάνουν κάτι, θα πρέπει τουλάχιστον να ξέρουν πώς, ποιο είναι το σωστό όνομα. Και αυτό δεν έγινε μία φορά, έγινε επανειλημμένος. Και μάλιστα σε μία συγκεκριμένη περίπτωση κάποιος που είχε ε, ε, πάρει τον τηλεφώνα του στο Clunking Bag για 70 χρόνια η πρώτη φορά που έμαθε για την οδηγία και την απαγόρευση να παίρνει τον τηλεφώνα ήταν από έναν αστυνομικό που τον έπιασε στον νόμο και του είπε ότι αν συνεχίσει να κάνει εξαγωγή από τον τηλεφώνα θα τον συνελάμβαναν και μάλιστα θα μπορούσε ε, να κληθεί να πληρώσει 500 εκατομμύρια πρόστιμο και να υποστεί και τρία χρόνια φυλάκιση. Άρα Φαντάζομαι συμφωνείτε ότι η επικοινωνία ήταν προβληματική. Γιατί λοιπόν δεν έχουμε καλή επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εύκολο να λέει κανείς να λέτε ότι εσείς φταίτε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έφταιγε η κυβέρνηση. Δεν έγινε διαβούλευση έγκαιρη. Οι διαβουλεύσεις που έγιναν είναι σαν αυτές ε, σε ε, στη σκοποβολή ε, τόσο γρήγορα. Πρώτα πετάτε το βέλος και μετά ε, το συζητάτε. Δεν έγινε λοιπόν ούτε διαβούλευση με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, ούτε ανάμεξή τους. Τίποτα δεν έγινε και μάλιστα αυτό που απαιτείται είναι ανάμεξη εμπλοκή και του Κοινοβουλίου. Έχουμε Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στην Ελλαδική Βουλή. Έπρεπε και αυτή να είχε αναμειχθεί. Δυστυχώ όλα έγιναν κατόπιν εορτή και μάλιστα ε, εμεί ήμασταν είτε στο Στρασβούργο είτε έγινε την εβδομάδα Επιτροπή. Οπότε ήταν πολύ ελληματική και προβληματική επικοινωνία. Και επίση λόγω αυτή τη έλλειψη επικοινωνία. Ε, εγώ συζήτησα με, με ε, Ιρλανδούς που έπαιρναν τα καύσιμά τους από τυρφώνες και επειδή δεν ήξεραν αυτό το θέμα, ε, καταλήξαμε σε σύγκρουση μεταξύ των ε, γεωργών και των αστυνομικών που χρειάστηκε να πληστούν κιόλα γιατί φτάσαμε, ήρθα στα χέρια κάποιος που για χρόνια ολόκληρα πήγαινε στο συγκεκριμένο τυρφώνα, του απαγορεύθηκε η πρόσβαση. Και ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Αν θέλετε καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε τέτοιες διαδικασίες. Είναι σαν να προσπαθεί κανείς να τον α, θρέψει με το ζόρι. Θα πρέπει να είστε πιο διακριτικοί, πιο διπλωμάτες και να έχετε διαβουλεύσει και επικοινωνία. Εγώ είμαι χορτοφάγος βέβαια και θα πρέπει να ακούσουμε μερικές φορές ε, και τους ε, συμπολίτες μας. Μιλούμε για ε, απειλούμενα είδη και θέλουμε να είμαστε ευαίσθητοι και να λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο απειλούμενο είδος που είναι η ανθρωπότητα. ο άνθρωπος είναι απειλούμενο είδος δεν υπερβολή, είναι γεγονός. Και έχουμε μία, έναν οργανισμό προστασίας της ε, Άγρας Πανίδας και το έχουμε, το έχουμε μετονομάσει γιατί πραγματικά αν θέλετε βελτίωση το, της υλοποίησης των περιβαλλοντικών στόχων θα πρέπει να βελτιώσετε την επικοινωνία και τη διαβούλευση. Εκεί αποτύχατε. Στην Ιλανδία δίνουμε μόνο έμφαση στο περιβάλλον. Δεν σας λέω να δώσουμε λιγότερο έμφαση στο περιβάλλον, αλλά λέω να δώσουμε έμφαση και σε άλλα δικαιώματα, να λάβουμε υπόψη και τις κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού. Γιατί χωρίς τον πληθυσμό δεν θα έχουμε περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Για πολλά χρόνια σε μια περιοχή οι κτηνοτρόφοι θα να, να απομακρύνουν τα κοπάδια τους και τελικά για να προστατευτούν κάποια φυτά και τελικά μετά από ένα διάστημα χρειάστηκε να, ε, χρειάστηκε να επιστρέψουν τα κοπάδια τους γιατί χρειάστηκε να επανέλθουν στις περιοχές αυτές. Και αυτό γιατί δεν έγινε καλή επικοινωνία από την αρχή. Στην Αλία το ίδιο. Έχουμε ένα οριζόντιο πρόβλημα. Και πολλοί γεωργοί στις παράκτιες περιοχές είναι και εραστέχνες αλής, αλής μικρής κλίμακας. Θα πρέπει λοιπόν να τους εμπλέξουμε και αυτούς ε, στα προγράμματα. Η επικοινωνία θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν πρώτα απ' όλα. Γιατί η ιδέα ότι ο η λέξη περιβαλλοντολόγος ή ε, οικολόγος έχει αρχίσει και ακούγεται σαν βρισιά, είναι πραγματικά τρομοκτικό. Αλλά εκεί καταντήσαμε επειδή δεν είχαμε εγκαίρους διαβουλεύσει και επικοινωνία. Συμφωνώ με τους στόχους της οδηγίας για τα διατήματα των πτηνών, αλλά πρέπει να μιλάτε στον κόσμο, να, έχετε, να λαμβάνετε τη γνώμη τους, γιατί δυστυχώς αρχίζουν οι άνθρωποι να σπανίζουν και αν εξαφανιστούν οι άνθρωποι ποιος θα διαχειριστεί τα χωράφια, εσείς θα πάτε να τα καλλιεργήσετε. Οι τεχνοκράτες, οι γραφειοκράτες, όχι. Εμείς θα πρέπει να το κάνουμε. Γι' αυτό αν δεν μας έχετε συμμάχους, μην περιμένετε να υλοποιήσετε όλους αυτούς τους στόχους. Πρέπει να βελτιώσετε την επικοινωνία μαζί μας. Ευχαριστώ. Κυρία Άουκεν, εγώ θα τα πω στα δανέζικα. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την πλήρη παρουσίαση και για την κάλυψη όλων των ερωτήσεων. Το πρόβλημα όμως είναι το ότι δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση αρκετά σοβαρά. Το θέμα είναι αν πιάνουν τόπο τα χρήματα τα οποία τίθενται για το Natura 2000. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό. Και μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι αυτό το ανέδειξε ως πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πολωνία. Γι' αυτό το πολωνικό δάσος. Όμως, αυτά εκ των υστέρων, γιατί μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή στην Ευρώπη δεν τηρείται η κοινωτική νομοθεσία. Οπότε χρειάζεται εφαρμογή της νομοθεσίας και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όποτε έχουμε παραβίαση του δικαίου. Χρειάζεται βέβαια και επαρκής χρηματοδότηση. Η ΚΑΠ απορροφά πάρα πολλούς πόρους. Θα πρέπει όμως να καθοριστεί ότι όλα αυτά τα χρήματα θα κατευθυνθούν προς την υποστήριξη της βιοποικιλότητας. Είδατε τι γίνεται με τα πτηνά σε γεωργικές ε, γέες. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο άσχημη είναι η κατάσταση. Να είδατε με τα κοτσίφια εξαφανίστηκαν. Άρα θα πρέπει και η βιοπικιλότητα να καλυφθεί από τις κοινωνικές πολιτικές, όπως και έχει τονιστεί τόσες φορές. Ε, αυτό είναι αναγκαιότητα. Όπως επίσης και για το θέμα των λίγων. Κάποτε όλα αυτά ήταν αυτονόητα. Κάποτε δεν τους κυνηγούσαμε και τώρα πληρώνουμε για να τους προστατεύουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το σύνολο του τοπίου και την οικονομική πτυχή και την αλλαγή του κλίματος. Χαίρομαι για όσα θέματα επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι βελτιώνεται η στάση μας σε σχέση με τα το πρόσφατο παρελθόν τέλο πάντων. Πάντω νομίζω ότι την εργαλειοθήκη, τα, τα μέσα, τα κατάλληλα τα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι να θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Ευχαριστώ. Άλλο θέλει το λόγο, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κ. Ντόφμαν. Δυστυχώ έφυγε. έχουμε αυτή τη συζήτηση με τους λύκους ε, και στη Γερμανία και λένε συνέχεια ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν περιοχές Natura 2000 που μας εμποδίζουν. Έχουμε κάποια είδη βεβαίως τα οποία πολλαπλασιάζονται πραγματικά αλματοδός, αλλά πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα. Υπήρχαν δηλαδή κάποια είδη βιτρίνας θα έλεγα, που πολλαπλασιάζονται καλά, αλλά από την άλλη πλευρά δεν ναι, βλέπουμε τη μεγάλη μείωση της βιοποικιλότητας ε, ειδών στο γεωργικό τοπίο. Εκεί πρέπει να παλέψουμε. Και έχουμε μια έρευνα στη δικιά μου την περιφέρεια. Είχαμε 95% ε, τη άγρια φαγκόγοτας εξαφανίστηκαν. Διάφορα είδη δηλαδή που απειλούνται. Αλλά όλος ο κόσμος μιλάει για τους λύκου μόνο. Τους κάστορες, ε, διάφορα ψάρια και τα άλλα προβλήματα δεν μας απασχολούν καθόλου. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε ψηφοφορία για τις περιοχές ε, οικολογικής προτεραιότητας. Πολύ σημαντική ε, συζήτηση για το ότι πράγματι ε, αν θα επιτραπεί η γεωργία σε 5% των περιοχών αυτών, αν θα χρησιμοποιηθούν ε, χημικά λιπάσματα. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτρέψει την χρήση χημικών λιπασμάτων εκεί πέρα, σε τόσο μικρές εκτάσεις πραγματικά είναι κρίμα. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση που θα αφορά γενικότερα τη γεωργική πολιτική, γιατί εκεί είναι τα σοβαρά προβλήματα. Και είναι πολύ σοβαρά τώρα από ό,τι στα... στις περιοχές που αναφέραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος τον λόγο, να επανέλθω στον κύριο Ντελγκάντο Ρόζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τα σχόλια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι κανείς δεν είναι κατά του σχεδίου δράση για τη φύση. Να πω το εξής. Λοιπόν, πρώτα προς τον κύριο Φλόρεντς. Ε, σεβόμαστε την κατάσταση των ε, γεωργών. Ξέρουμε πόσο σκληρά περνάμε. Βεβαίω οι χαμηλέ τιμέ δεν έχουν σχέση με την Natura 2000, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στο παρελθόν ε, ε, και τώρα ε, θεωρούν ότι δεν τους έφταναν όλα τα άλλα, έχουν και την Natura 2000 στο κεφάλι τους. Μα αναφερθήκατε στους κορμοράνους. Το ίδιο ισχύει και για τους κάστορες ε, και άλλα είδη. Δηλαδή, αν ε, προκάλεσαν κάπου καταστροφές όπως αναφέρεται, ε, τότε ξεκαθαρίζουμε το ότι ε, πρέπει να γίνει. Επίσης ε, κάποια είδη είναι προστατευόμενα, κορμοράνι κτλ. Οπότε υπάρχουν παρεκκλήσεις για να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον όπως η αλληλεία, αλλά εγώ θα έλεγα το εξής. Ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το ότι δείγμα δεν σημαίνει ότι πρέπει να προστατευτεί κάποιο συγκεκριμένο δείγμα για να προστατευτεί ένα είδος. Ε, υπάρχει, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Υπάρχει όμως μια κακή πρακτική που ακολουθείται παντού, η οποία είναι «Α, φταίνει οι Βρυξέλλες». για πολλά πράγματα φταίει η Κομισιόν και η νομοθεσία, αλλά η διαχείριση και οι εξαιρεσει είναι περιφερειακό και εθνικό θέμα, δεν είναι κάτι που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Βεβαίως, ε, έχουμε λόγο σε κάποια πράγματα, ε, αναφέρθηκαν οι Σουηδικοί λύκοι. Αλλά βεβαίω ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο βιώσιμο πληθυσμό είναι ο αριθμό χ, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και την γενετική ανθεκτικότητα στη Σουηδία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ενδογαμίας που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οπότε συζητάμε με τις Σουηδικές αρχές. Οπότε πράγματι πρέπει να συζητήσουμε και με τους αγρότες άμεσα που πρέπει να έχουν ένα βιώσιμο εισόδημα, αλλά θα πρέπει να έχουν βεβαίως και μια αποζημίωση ε, τώρα, αποζημίωση είναι για διαφυγόντα εισοδήματα από το Natura 2000. Πράγματι, είναι ενσωματωμένο αυτό το ότι πράγματι οι αγρότες πρέπει να μπορούν να βγάζουν τα προστοζήν και είναι ενσωματωμένο στο πρόγραμμα. Τώρα, για το ζήτημα της ευελιξίας στα χαρτιά. Γι' αυτό ακριβώς ε, το σχέδιο δράσης αυτό χρειάζεται. Γιατί εμείς ακριβώς έχουμε το χαρτί, το πνεύμα και το γράμμα των οδηγιών είναι ευέλικτο αν το διαβάσετε και γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις ε, όπου είχαμε αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Φλανάγκαν, όπου είχαμε μηδενική ευελιξία, είχαμε κακές πρακτικές, αλλά είχαμε και ορθές πρακτικές. Για το θέμα τώρα των ε, ανθρώπων και των επιβλαβών ειδών, ποντίκια, αλίκη κτλ. Οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τα ποντίκια και τους λύκους με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που αγαπάν τους λύκους, κάποιοι δεν έχουν αντίληψη του τι προκαλεί ο λύκος ε, στις αγροτικές κοινότητες. Οπότε ε, μπορούμε να αναφέρουμε πολλές επιτυχημένες ιστορίες στην Ευρώπη. Κάποιες πρακτικές χάθηκαν. Ε, πρέπει λοιπόν να βρεθεί η σωστή ισορροπία και όχι εις βάρος του ζωικού κεφαλαίου και των αγροτών. Για να βρούμε λοιπόν αυτή την ισορροπία. Οι ηλίκοι παίζουν έναν οικολογικό ρόλο. Όχι, δεν πάει έτσι. Το οικοσύστημα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Εγώ δεν έχω πληροφορίες περί υβριδικών ειδών ε, με, τους... Ε, σκύλους. Υπάρχει βεβαίως, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κίνδυνος να αντικατασταθούν πλήρως οι λύκοι. Ε, το θέμα της επικονίασης ε, της κυρίας Κάντενμπαχ. Εμείς θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το ζήτημα της επικονίασης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ανέφερε η κυρία Κάντενμπαχ Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις όπου αυτό ισχύει σωστά, αλλά υπάρχουν και πολλές κακές πρακτικές. Πρέπει να δούμε τις σωστές πρακτικές και να τις εναρμονίσουμε. Να δούμε και τον διμερή ε, διάλογο και το τι θα φέρει. Ε, χαίρομαι λοιπόν επίσης ε, κυρία σμάκερ ε, για τις υψηλές ε, προσδοκίες, αλλά δεν αρκεί μόνο να, υπάρχει, να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές σε ένα site στα αγγλικά, πρέπει να είναι σε όλες τις γλώσσες και οι εθνικές αρχές να τις διαδώσουν. Το θέμα τώρα των στόχων 2020 ε, για τη βιοπικιλότητα. Ναι, γιατί μέχρι το 2020 είναι οι στόχοι, δεν τους έχουμε επιτύχει, το σχέδιο δράσης βοηθάει, αλλά θα έλεγα δύο πράγματα. Πρώτον, οι πράσινες υποδομές είναι μια συνεισφορά που πάει πέρα από το δίκτυο Natura 2000. Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι αρκετά χρήσιμο. Οι κατευθύνες γραμμές για το πώς θα λάβουμε υπόψη τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Γιατί εάν σε όλους τους τομείς ε, λαμβάνεται αυτό υπόψη, σε όλα τα, όπως κάνουν κάποιες χώρες ε, στην εθνική του νομοθεσία, αυτό μπορεί να κάνει πολλά για να υπάρξει ακριβώς αυτή η αλλαγή στην κοινωνία για να προστατευτεί η ιδιοποικιλότητα. Τώρα, μετά το 2020 είναι ένα αυτό θέμα όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για τον κόσμο. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι έχουμε κάποιους ε, στόχους ε, που θα πρέπει να επιτύχουμε. Μάλλον δεν θα τους πετύχουμε όλοι, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα επιτύχουμε μια παγκόσμια στρατηγική μετά το 2020 που δεν θα επαναλαμβάνει απλά κάποιους στόχους. Ε, και το προσέχουμε αυτό. Κύριε Φλάναγκαν. Μάλιστα. Ε, πολύ παραστατικό το παράδειγμα που μας δώσετε για το τι πρέπει να αποφύγουμε. Σίγουρα δεν είναι αυτή η καλύτερη προσέγγιση για τους αγροκτήμα, αγροκτήμονες και γεωκτήμονες. Και μάλιστα μετά το Natura 2000 έπρεπε να τους συγχαρούμε ε, για αυτό που έκαναν. Αλλά μετά, λόγω των περιορισμών, ε, έχουν την αίσθηση ότι τους δέσαμε τα χέρια. Σίγουρα έτσι δημιουργείται μια έξαρση της καχυποψίας και της δυσπιστίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε πολλές χώρες βελτιώθηκε αυτή η κατάσταση της δυσπιστίας, γιατί το, ο ξεματόχος που ήταν αρμόδιος για την επαφή με τους τοπικούς ε, φορείς πραγματικά κατάφερε και άλλαξε αυτό το κλίμα και το έκανε πιο θετικό. Βέβαια, σε μερικέ περιπτώσει θα χρειαστεί περισσότερη προστασία, αλλά είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε εμπλοκή και ανάμειξη των τοπικών φορέων και των γεωργών. Φυσικά δεν μπορούμε να πάμε στο κάθε χωριό και σε κάθε κομμόπολη, δεν έχουμε αρκετό προσωπικό, αλλά θέλουμε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και του τοπικού και περιφερειακού φορεί. Γι' αυτό και τόνισα πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με τη με την Επιτροπή Περιφερειών και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξεκινήσουμε ένα γνήσιο διάλογο και να οικοδομήσουμε αυτή την χαμένη εμπιστοσύνη και να εξασφαλίσουμε τις συνέργειες ε, και με τους οικολόγους και με τους ε, γεωργούς. Ε, δεν είχαμε παντού αποτυχίες, μερικές φορές είχαμε και επιτυχίες ευτυχώς, αλλά, αλλά σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κύριε Άουγκεν, θέλουμε προσοχή στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης και επίσης ε, στη μελλοντική ΚΑΠΑ να προσέξουμε το θέμα της προσημείωσης των κονδύλιων. Το λέμε αυτό και στο τωρινό σχέδιο ε, δράσης και στην τωρινή ΚΑΠ. Επίσης, το θέμα του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών, άλλο σημαντικό θέμα που μας ενδιαφέρει και στα οδηγίε για τη φύση και στο Natura 2000. Κύριε Χόισλινγκ, πολύ σωστά είπατε ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα ε, είδη που ε, εξαπλώνονται και πολλαπλασιάζονται. Όμως μερικά δυστυχώς μειώνονται. Και το παρατηρούμε αυτό. Και το Natura 2000 δεν λύνει το πρόβλημα παντού, αλλά προσπαθεί να αναχαιτήσει αυτή, αυτή την απειλή ή να βελτιώσει την κατάσταση της διατήρησης σε πολλά είδη. Σε ευχαριστώ ε, για την υποστήριξή σας ό,τι αφορά την απαγόρευση χρήση φυτοφαρμάκων στις περιοχές οικολογικής εστίασης. Σίγουρα επειδή σε τέτοιε περιοχέ οικολογική αιστεία θέλουμε να τονώσουμε τη βιοπικιλότητα, καλό είναι να απαγορεύουμε τα φυτοφάρμακα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους συνάδελφου που έλαβαν μέρος στη συζήτηση και κυρίω τον κύριο Νταλκάδο Ρώσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ήταν και το τελευταίο σημείο της ημερήσια διάταξη, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μόνο διάφορα μας έμειναν, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία ούτως ή άλλως. Δεν, έχουμε χρόνο, αλλά μπορείτε και να στείλετε την ερώτηση στην Επιτροπή. Εκτός μικροφώνου δυστυχώς ο κ. Φλάναγκαν. Anyway, so uh, our next is going to be... Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα και η επόμενη τακτική συνεδρίαση στις Βρυξέλλες 21 και 22 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ και καλό μεσημέρι.